Καλησπέρα σε όλους, αν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα με το χρόνο. Και ξέρετε, όταν ε, μας ξεφεύγει ο χρόνος, έχουμε και τη σχετική εμπειρία, ξέρετε τι συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη δημόσια κρίση για την κοινή οργάνωση αγορά ε, για τα αλληλευτικά προϊόντα και τα προϊόντα δεδοκαλλιέργεια στο πλαίσιο τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική Πολιτική ε, με Ε, και θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τους προσκεκλημένους που θα συμμετάσχουν στην εδρίαση αυτή, την οποία την έχουμε διαιρέσει σε δύο μέρη και καταρχήν ε, θα λάβουν το λόγο οι κύριοι Γιάννα Μασουίν, Πιμ Βίσερ και Χωσέ Απολινάριο και στη συνέχεια στο δεύτερο πάνελ θα πάρουν το λόγο η κύριοι Τόρσεν Μάρτισον, η κυρία Γκέρλινγκ και ο κύριος Φερνάντες. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, μου να, πριν ξεκινήσουμε να πω το εξή, ότι μου είπαν ότι η κυρία Γκέρλινγκ ίσως ε, θα μπορούσε να πάρει πρώτα το λόγο, αν δεν υπάρχει αντίρρηση από τον κύριο Τόρσεν, να αλλάξουμε τη σειρά. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Και χωρίς κοινοτριβή θέλω να σας καλωσορίσω εδώ στο Κοινοβούλιο σε μια σημαντική συγκυρία. Συζητάμε τη μεταρρυθμίση της κοινής ελευτικής πολιτικής ε, και πιστεύω ότι αυτή η δημόσια ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν έχουμε αθρώα προασέλευση βέβαια, αλλά υπάρχει αρκετή ποιότητα. Έτσι λοιπόν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή τη σκοπιά. Και θα δώσω το λόγο στον συγκητή, στον κύριο Στίβενσον, για να κάνει μια σύντομη εισαγωγή και στη συνέχεια, με τη σειρά που ανέφερα, θα πάρουν το λόγο οι προσκεκλημένοι μας. Θέλω να παρακαλέσω τους προσκεκλημένους γιατί Έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσπαθείτε, να προσπαθήσετε να σεβαστείτε τα 10 λεπτά που έχουν προβλεφθεί για την παρέμβασή σας για να κάνουμε και μια συζήτηση στη συνέχεια με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και να θέσουμε τις ερωτήσεις και να έχουμε και ένα διάλογο. Έχετε το λόγο κύριε Στίβενσον. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους ομιλητές ε, που έχουν ε, έρθει από μακριά για να συμμετάσχουν σήμερα στην ε, ακρόαση αυτή. Εγώ είμαι εισηγητής για την κοινή οργάνωση αγοράς και για μένα είναι σημαντικό το θέμα. Εκτιμώ πολύ την συμβολή των εμπειρογνωμόνων του τομέα. Και γι' αυτό θα είμαι σύντομος Όλοι λάβατε νομίζω το πρώτο έγγραφο εργασίας μου, το οποίο ήταν κάπως πιο ογκώδες, το οποίο μεταφράστηκε σε όλες τις ε, γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω επίσης ότι έχετε στο φάκελό σας το πιο σύντομο δεύτερο έγγραφο, το οποίο έχει, στόχο, ε, το οποίο έχει τίτλο «Στόχοι», «Objectives», το οποίο ε, περιγράφει την κατεύθυνση προς την οποία προβλέπω να πάει η έκθεση. Στην Επιτροπή μας χθε είχαμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Συμμετείχαν σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και για αυτούς, ε, αν όχι για τους υπόλοιπους, ε, θέλω να είμαι σύντομος και να δώσω περισσότερο χρόνο στους επιρογνώμονες. Η βασική αρχή πίσω από την έκθεση για την κοινή οργάνωση αγορά που αποτελεί μία από τι τρει νομοθετικέ εκθέσει για την μεταρρύθμιση τη κοινή αλλιευτική πολιτική είναι το μέλλον της αγοράς στην Ευρώπη, οι οργανώσει παραγωγών στην Ευρώπη και υπάρχουν 214 τέτοιε, και μάλιστα πολλές από αυτές είναι σκεντρωμένε σε ένα-δύο κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη όπως η Ιρλανδία ή κάτω χώρες έχουν πολύ λίγες οργανώσεις παραγωγών, ενώ ε, κράτη-μέλη όπως η Ισπανία έχουν πολύ μεγάλο αριθμό. Και μερικές από αυτές τις οργανώσεις έχουν ε, ιστορία δεκαετιών. Όλες παίζουν ε, λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο, ζωτικό ρόλο στο μέλλον, των... στο μέλλον της αλληλείας μας. Η έκθεση λοιπόν για την κοινή οργάνωση αγοράς εξετάζει το πώς μπορεί να συντονιστεί ο ρόλος τους πώς μπορούν να εξεταστούν οι διακλαδικές οργανώσεις, οι διεθνικές οργανώσεις, πώς μπορούμε για όλους, για τους αλληλείς, για τους μεταποιητές, για τους ε, ε, ε, ιδιοκτήτες των σκαφών, για τους καταναλωτές, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αγορά προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Από τα έγγραφα που έχω υποβάλει θα έχετε δει κάποιες από τις ιδέες που έχω υποβάλει για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Και θα είδατε και την επικάλυψη ανάμεσα στην έκθεσή μου και την ε, βασική μεταρρύθμιση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής όπως, ε, σε τομείς όπως είναι οι μεταβάσιμες ε, αλλιευτικές παραχωρήσεις, σε τομείς όπως είναι η περιφερειοποίηση ή οι απορρίψεις, διότι οι οργανώσεις παραγωγών θα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο ε, κατά τη διαχείριση της αλληλείας ε, ε, στην καθημερινή ζωή όσον αφορά τα ΤΑΚ, τον περιορισμό της αλληλευτικής προσπάθειας. Στα θέματα αυτά θα ήθελα να δω πιο ισχυρό ρόλο των οργανώσεων παραγωγών και νομίζω ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή μας θέλουμε να δούμε μια λογική περιφερειοποίηση που θα επιτρέψει στους οργανώσεις παραγωγών να παίξουν αυτόν τον πιο σημαντικό ρόλο μαζί με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις απορρίψεις, η πρόταση της Επιτροπής ε, προτείνει οι οργανώσεις παραγωγών να παίξουν ρόλο κλειδί. Όλα αυτά τα ψάρια τα οποία ε, λογικά απορρίπτονται νεκρά στην ε, θάλασσα, αυτά να ε, εκφορτώνονται μετά από απαγόρευση βαθμιαία ε, τουλάχιστον ε, για κάποια είδη. Η Κομισιόν προτείνει τα ψάρια αυτά να διανεμηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε γυροκομεία και άλλα ιδρύματα. Ε, μαζί με τις ε, οργανώσεις παραγωγών σε όλη την Ευρώπη πιστεύω ότι αυτό είναι ανόητο. Όχι μόνο θα υπονομεύσει την αγορά, διότι αν αρχίσει κανείς να χαρίζει ψάρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα σταματήσουν να τα αγοράζουν. Πέρα από αυτό όμως, ποιος θα πληρώσει τις οργανώσεις παραγωγών για την μεταποίηση αυτών των απορρίψεων. Ε, 1,4 ε, εκατομμύρια τόνοι περιμένουμε να μεταποιηθούν από τις οργανώσεις παραγωγών χωρίς καμία αποζημίωση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ε, εξαλείψουμε τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα με τεχνικά μέσα. Και αυτό πρόκειται για τροποποίηση του βασικού κανονισμού. Θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των ψαριών που θα αποτελούσαν αντικείμενο απόρριψης με τη χρήση τεχνικών μέτρων και κατόπιν θα πρέπει να βρούμε λογικό τρόπο διάθεσης των ηχθείων αυτών που υποχρεωτικά εκφορτώνονται είτε για την παραγωγή ηχθιάλευρου και ηχθιέλεου, ε, για την μεταποίηση ε, για ε, ηχθιοτροφέ ή για άλλους λόγους. Θα πρέπει να είμαστε ε, ε, ευέλικτοι όσον αφορά το πώς θα γίνει αυτό και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι αλληλείς ώστε να συμμορφώνονται με αυτούς τους νέους κανονισμούς. Όσον αφορά το έγγραφό μου που περιγράφει τους στόχους, ε, θα ήθελα να αναφέρω και το όραμά μου για την επόμενη δεκαετία. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αγορά για όλους, για τους μεταποιητές, για τους αλληλείς, για τους ε, δημοπράτες. Ε, ήδη έχουμε ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίων, ε, έχουμε παρακολούθηση των πλοίων με δορυφόρο. Στην Γαλλικία έχουν μια τεχνολογία με μαγνητική κάρτα στην, στην προβλήτα στο λιμάνι. Θα πρέπει όλοι οι καπετάνοι, να, όλοι οι κυβερνήτες πλοίων να συμμορφώνονται με αυτό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε να αυξηθούν οι τιμές ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν ε, καλής ποιότητας υγιεινά τρόφιμα και έτσι περνάω στο επόμενο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, την επισήμανση που παίζει σημαντικό ρόλο στην έκθεσή μου επίσης. Υπάρχουν κάποιες διαμάχες σχετικά με το τι θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνεται στην ετικέτα, στην επισήμανση. Ε, πέρσι είχαμε στο Κοινοβούλιο τριμερή διάλογο που αφορούσε την ενημέρωση των καταναλωτών. Πολλές οργανώσεις παραγωγών μου είπαν ότι αφού περάσαμε αυτήν την βασανιστική διαδικασία ε, για να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να υπάρχει στην επισήμανση όλων των τροφίμων, τώρα έχουμε νέες προτάσεις της Κομισιόν για νέα επισήμανση στα προϊόντα αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Και για το θέμα αυτό λοιπόν ε, κάνω κάποιες προτάσεις. Η θεοκαλλιέργεια έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον ε, στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Η Κομισιόν το αναγνωρίζει το γεγονός αυτό. Επίσης προτείνει να, υπάρξουν περιφερειακά, να, υπάρξει, να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό συμβούλιο για την ηχθειοκαλλιέργεια. Ε, ο τομέας της ηχθειοκαλλιέργειας έχει δείξει πολύ ενθουσιασμό για το θέμα αυτό και στο έγγραφό μου με τους στόχους, ε, με τον τίτλο Objectives, ε, αναφέρονται ε, σχετικές συστάσεις. Μετά την σύντομη αυτή εισαγωγή, θα ήθελα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Να περάσουμε στους εμπειρογνώμονες. Καταρχήν έχει το λόγο ο κύριος Ιαν Μαξουίν. Uh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μου δίνει για μας που εκπροσωπούμε τον κλάδο να απευθυνθούμε σε, μας, σε εσάς. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτό της διαδικασίας μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όσον αφορά πολλούς από εμά που εκπροσωπούμε τον κλάδο, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι η μεταρρύθμιση του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με την γενικότερη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Για πάρα πολύ καιρό η κοινή οργάνωση αγοράς θεωρείται ως ξεχωριστή πολιτική που είχε ελάχιστη σχέση με τις γενικότερες πτυχές πολιτικής στον τομέα της αλίας. Η κοινή οργάνωση αγοράς πρέπει και μπορεί να συμβάλλει προς, τους γενικότερους, προς την επίτευξη των γενικότερων στόχων της κοινή ελευτικής πολιτικής. Θα ήθελα σύντομα, σήμερα το απόγευμα, είναι να αναφερθώ στην κοινή οργάνωση αγοράς και να την τοποθετήσω στο γενικότερο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Γιατί πιστεύω ότι στο παρελθόν ένας από τους βασικούς λόγους εσφαλμένων πρακτικών που βλέπαμε στον κλάδο, όπως για παράδειγμα οι εκφορτώσεις άνω των ποσοστώσεων και οι απορρίψεις, ήταν οι χαμηλές τιμές. Οι χαμηλές τιμές δημιουργούν ένα κίνητρο για τους αλείς, προκειμένου να προχωρούν σε εκφορτώσεις άνω των επιτρεπόμενων ποσοστώσεων, και κατά αυτόν τον τρόπο υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Οι χαμηλέ τιμέ δημιουργούν τελικά ένα κίνητρο για μεγαλύτερη αλίευση. Η βιολογική βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα όταν συνοδεύεται από την οικονομική βιωσιμότητα. Η οικονομικά ασύμφορη αλία είναι πολύ πιο πιθανό να είναι και μη βιώσιμη από βιολογικής πλευράς, καθότι ασκείται μεγαλύτερη πίεση για υπεραλίευση και για εκφορτώσεις άνω των επιτρεπόμενων ορίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η κοινή οργάνωση αγοράς να μας επιτρέψει να επιτέχουμε τον στόχο μιας οικονομικά συμφέρουσας αλίας και κύριε Πρόεδρε αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του μηχανισμού τιμών. Οι ελευτικές εταιρείε είναι γενικά μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Οι εταιρείε μεταποίηση όμω από την άλλη είναι συνήθω αρκετά μεγάλε, μόνο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ανάλογα με το είδο ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Σε ορισμένε χώρε, οι πολιτέ είναι ιδιαίτερα δυνατοί και έχουν πολύ δυναμική παρουσία στην αγορά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να θέτουν τι τιμέ σε επίπεδα που είναι οικονομικά ασύμφορα για του αλείς. Και ακριβώ για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν οι οργανώσεις παραγωγών ήταν ουσιαστικά μία απόπειρα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μία αντισταθμιστική μονοπωλιακή εξουσία σε ένα κλάδο όπου ο μεμονωμένος τελικό, τελικά αλλιεύς μπορεί να, να μειωθεί σε έναν άτομο που απλώς αποδέχεται τις τιμέ που του επιβάλλονται εκ των άνω. Οι οργανώσεις παραγωγού λοιπόν θέλανε να εξασφαλίσουν ρεαλιστικές τιμές για τα αλλιεύματα των ψαράδων και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει ποτέ να επιτύχει τον στόχο της βιώσιμης αλίας αν η αλία δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η διαδικασία μεταρρύθμισης και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η πρόταση για την απόσυρση του συστήματος παρέμβασης δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το σύστημα τιμής απόσυρσης αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας για τους ελευτικούς στόλους. Το επιχείρημα ότι οι δαπάνες για τα αποσυρώμενα από την αγορά λιεύματα είναι πολύ χαμηλές ουσιαστικά είναι ανεφουσίας. Στην πραγματικότητα καταδεικνύει ότι το σύστημα τελικά λειτουργεί στην πράξη. Το εφιστάμενο σύστημα θέτει ένα κατόφλι στην αγορά, το οποίο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της αγοράς. Αν όμως καταργήσουμε το κατόφλι αυτό, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο τομέας της μεταποίησης θα εξαναγκαστεί από τους λιανοπολιτές να μειώσει τις τιμές. Και ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία λέγονται για την ιχνηλασιμότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα, ο βασικός καθοριστικός παράγοντας αγοράς αλλιευμάτων από το καταναλωτή παραμένει ένας, η τιμή. Και αυτό καταδεικνύεται ξεκάθαρα την, στην παρούσα περίσταση με τον Σολομό το κλείσιμο ενό μεγάλου μέρους της παραγωγής Σολομού από τη Χιλή και η μεταστροφή των Ευρωπαίων παραγωγών προς τη Βόρεια Αμερική σε μια πολύ σημαντική αύξηση της τιμής του Σολομού. Η αντίδραση στην αύξηση αυτή ήταν τελικά μία μείωση της κατανάλωσης και το τελικό αποτέλεσμα είναι τελικά η πρώην τιμή Σολομού εκτροφής να είναι περίπου 50% από αυτό που ήταν πριν από ένα χρόνο με τις αυξήσεις που έχουμε στο Γάδο και στον Εγκλεφίνο, στη θάλασσα του Μπάρεντς και στην Ισλανδία, η τιμή του κορέγονου, του ασπρόψαρου, θα μπορούσε να κατακαιρματιστεί αν δεν υπήρχε ένα απαραίτητο κατόφλι στην αγορά. Ήδη βλέπουμε πολύ σημαντική μείωση στις τιμές όσον αφορά τον γάδο από την Ορβηγία και τη Ρωσία. Αν μειωθούν όμως οι τιμές, τότε και οι βιώσιμες πρακτικές θα εξαφανιστούν καθώς θα προσπαθούν οι αλλοίς να επιζήσουν. Το επιχείρημα λοιπόν ότι από μόνη τη η αγορά θα πρέπει να καθορίσει τις τιμές μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά τελικά δεν λαμβάνει υπόψη του κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η παραγωγή στον ελευτικό τομέα έχει μια συγκεκριμένη οροφή, την οροφή των ποσοστώσεων. Επομένως η φυσιολογική αντίδραση στη μείωση των τιμών, δηλαδή μια αύξηση της παραγωγής, δεν μπορεί να συμβεί στην πράξη. Η εγχώρια αγορά λοιπόν της αλίας έχει μια συγκεκριμένη οροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απορρέει από το σύστημα των ποσοστώσεων. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να εξεταστεί από κοινού μαζί με τις πάρα πολύ μεγάλες προμήθειες κορεγόνου, οι οποίες φτάνουν τελευταίο καιρό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιχείρημα ότι δεν θα πρέπει να καταναλώνουμε τα χρήματα των φορολογούμενων για την καταστροφή των τροφίμων, ουσιαστικά Προφανώ ισχύει και είναι αποδεκτό. Αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι αυτοί περιέργω σιωπούν κάθε φορά που πρέπει να πληρώσουν παραγωγού για να παράγουν ζυζάνια αντί για να καλλιεργούν τρόφιμα. Το σύστημα απόσυρση το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή δεν οδηγεί σε μια καταστροφή των τροφίμων. Οι αποσυρθέντες ηχθείς ουσιαστικά γίνονται ηχθιέλαια και ηχθιάλευρα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές στο σύστημα της ιδετοκαλλιέργειας και αποτελούν επίσης μια πολύ σημαντική πηγή πρωτεϊνών και ω3 για τον διατροφικό τομέα. Επομένω, η μεταρρυθμισμένη κοινή οργάνωση αγορά θα πρέπει να επιτρέπει την παρέμβαση για την κατανάλωση που δεν προορίζεται για τον άνθρωπο. Από τότε που δημιουργήθηκε η κοινή οργάνωση αγορά, το σύστημα παρέμβασης με το σύστημα τιμών απόσυρση έχει δραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της αλεία και, έχει, και υπάρχουν πάρα πολλέ θέσει εργασία που συνδέονται με το σύστημα αυτό. Αν δεν υπήρχε το σύστημα παρέμβαση, κυρίε και κύριοι, θα έχουμε ένα πραγματικό κίνδυνο να πέσουν οι τιμέ κάτω από το επιτρεπτό επίπεδο. Από το επίπεδο δηλαδή αυτό που μα επιτρέπει να έχουμε μια οικονομικά συμφέρουσα και βιώσιμη αλία, ιδίω για μια αλία μικρή κλίμακα παράκτια. Οι οργανώσει παραγωγών μπορούν να δραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση τη αλεία, καθώ επίση και στην διάθεση στην αγορά των αλλιευμάτων. Οι προτάσει όμω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί η αγορά ω μέσο για να ελεγχθούν οι απορρίψει δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Η όλη έννοια ότι τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα θα πρέπει να εκφορτώνονται και στη συνέχεια να καταψύχονται προτού δοθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσει και το καθεξής δεν είναι καθόλου λογική. Καταρχάς, θα είχαμε πολύ σημαντικέ δαπάνε μόνο και μόνο από τη διαδικασία κατάψυξη αυτών των εκφορτώσεων και η ποιότητα των μικρών ιδίω ψαριών επιδεινώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εγγυηθούμε την ποιότητα τέτοιων εκφορτώσεων, καθότι τα πληρώματα στα διάφορα σκάφη θα ενδιαφέρονται καταρχάς για τα πια οικονομικά συμφέροντα είδη και δεν θα ασχολούνται καθόλου με τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα. Και ποιο θα πληρώσει ακόμα και τον πάγο που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να, να τα καταψυχθούν εν πλώ τα αλλιεύματα αυτά και ποιο θα πληρώσει για τα τεράστια κοντέινερ που χρειάζονται και τη μεταφορά των ψαριών. Αλλά ακόμα και αν τα φέρουμε τα ψάρια αυτά στην ακτή, τα εκφορτώσουμε και τα καταψύχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία αγορά για τα αλλιεύματα αυτά σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Επομένως η λύση για τις απορρίψει βρίσκεται στο να μην αλλιεύονται καν τα ίδια αυτά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί για τα μικρά ψάρια μέσω κάποιων τεχνικών μέτρων. Το πραγματικό πρόβλημα όμως παραμένει στην απόρριψη των εμπορεύσιμων ψαριών. Και θα έλεγα ότι η λύση για αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στα επίπεδα που θέτουμε στα πλαίσια των συνολικών επιτρεπόμενων αλλιευμάτων. Το να θέτουμε τάξ για συγκεκριμένα είδη και να χρησιμοποιούμε τα τάκ αυτά για πάρα πολλά είδη στη συνέχεια θα είναι ένας τρόπος για να καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα της απόρριψης των εμπορεύσιμων ψαριών. Πρέπει να έχουμε ένα γενικότερο σύστημα και να μην έχουμε απλώς συστήματα τα οποία απευθύνονται σε ειδικέ κατηγορίες ψαριών. Οι οργανώσει παραγωγών βρίσκονται στην καρδιά και τη κοινή οργάνωση αγορά. Θα πρέπει να έχουν όμω τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Η, η αναγνώριση των ομάδων παραγωγών θα πρέπει να, να γίνεται συστηματικά, να του θεωρούμε πραγματικού εταίρου, να έχουν την απαραίτητη παρουσία προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Χρειάζονται επίση απαραίτητε αρμοδιότητε για να, να πετύχουν του στόχου του. Η διαχείριση της αλίας είτε έχει να κάνει με τις προμήθειες είτε με τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων θα πρέπει να περνά και από τις ομάδες παραγωγών. Οι ομάδες παραγωγών θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ρυθμιστεί η δραστηριότητά τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να σταματάνε διάφορα σκάφη από το να αλλιεύουν προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη βιωσιμότητα. Θα πρέπει να μπορούν να ρυθμίζουν τις προμήθειες προϊόντων στην αγορά. Ο λιαυτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, περνάει πολύ δύσκολες ε, στιγμές. Οι δαπάνες του κλάδου αυτού έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από διάφορους παράγοντες όπως η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου. Επίσης, τα αποθέματα δεν βρίσκονται όλα στην καλύτερη δυνατή θέση, μολονότι έχουμε πολύ σημαντική ανάκτηση αποθεμάτων στη Βόρεια Θάλασσα και σε άλλες περιοχές. Και η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι είναι σε θέση να ρυθμίσει αυτή τη στιγμή τις προμήθειες που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι σίγουρο θα καταφέρει να το πετυχαίνει αυτό πάντα στο μέλλον. Επίσης, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ε, οι τιμές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις αγόμενες προμήθειες θα είναι πάντα πιο ανταγωνιστικές από αυτές που χρησιμοποιούνται για τις εγχώριες προμήθειες. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχει μια αυξανόμενη διεθν... ένας αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός για όλα τα προϊόντα και ιδίω όμως ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος για τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες όπως η Κίνα. Η ζήτηση για αλλιεύματα στην Κίνα έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και φαντάζομαι ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η διατροφική λοιπόν ασφάλεια, η επισητιστική μάλλον ασφάλεια είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλο και περισσότερο στο μέλλον. Το να καταφέρουμε να δώσουμε τα απαραίτητα τρόφιμα προς τους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί το να έχουμε μια πολύ, ένα πολύ καλό ελευτικό κλάδο. Αυτό σημαίνει όμως ότι ο ελευτικός στόλος και ο γενικότερος τομέας των θαλασσινών θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε ένα επικερδές και βιώσιμο περιβάλλον. Είναι λοιπόν θεμελιώδες η μεταρρυθμισμένη κοινή οργάνωση αγοράς να καταφέρει να συμβάλλει στη διαδικασία αυτή. Κύριε Πρόεδρε, μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα η εργασία που έχουμε δει να γίνεται μέχρι στιγμής από την Επιτροπή Αλίας. Από ό,τι φαίνεται και εσείς πιστεύετε τα ίδια πράγματα με μένα και πιστεύω ότι το γενικότερο πλαίσιο ανταλλαγή απόψεων το οποίο βλέπουμε να λαμβάνει η χώρα τελικά μας πείθει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε αμέσως ε, στο δεύτερο προσκεκλημένο μας, ε, τον κύριο Πινδίσερ. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανώσεων Παραγωγών. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σύντομα θα σας παρουσιάσω το περιεχόμενο της παρουσίασής μου. Θα σας παρουσιάσω την ΕΑΠΟ, την, ε, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων Παραγωγών. Ε, θα αναφερθώ στα βασικά στοιχεία στην διαδικασία αναθεώρησης και ε, νέα θέματα τα οποία θέλω να σας αναφέρω, τα οποία εν μέρη θα αποτελούν επανάληψη αυτών που μόλις ανέφερε ο κύριος Μαξουίν. Η ΕΑΠΟ είναι Πανευρωπαϊκή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών. Εκπροσωπούμε οργανώσεις παραγωγών από 10 κράτη-μέλη από τον βορρά στον νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα μέλη μας ε, εκπροσωπούν περίπου 10.000 σκάφη και 3,5 εκατομμύρια τόνων εκφορτώσεων στην ε, στον Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό με αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια. Εδώ βλέπετε ε, μια μικρή επισκόπηση του είδους των σκαφών που εκπροσωπούν ε, από μεγάλες τράτες μέχρι πιο μικρά σκάφη. Όλα αυτά ε, αντιπροσωπούνται από την Ένωσή μας. Εντός της ΕΑΠΟ Έχουμε συζητήσει την ε, μεταρρύθμιση εδώ και πολύ καιρό. Από το 2008 ξεκινήσαμε, καθότι τότε προβλεπόταν ξεχωριστή μεταρρύθμιση. Ε, μετά όμως ε, είδαμε ότι και ότι θα συνδυαστούν οι μεταρρυθμίσεις σε δύο διαφορετικούς τομείς. Είχαμε συζήτηση στην ΑΚΦΑ. Το... Η κυρία Δαμανάκη παρουσίασε τις προτάσεις της τον Ιούλιο και στο Εδιμβούργο ε, συζητήσαμε ε, την μεταρρύθμιση με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν σχηματίσαμε ομάδα εργασίας όπου συμμετείχαν μέλη της ε, Ένωσής μας και όλα αυτά ε, είχαν ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο θέσης του Ιανουαρίου 2012, το οποίο θα σας διανεμηθεί. Τα βασικά κλειδιά της παρούσας ε, ΚΟΜ είναι ότι είναι ειδικά πολύπλοκοι. Έτσι δυσκολεύονται οι εθνικές διοικήσεις να ασχοληθούν. Το κλειδί, όπως είπε ο κύριος Μασουίν, είναι ο μηχανισμός παρέμβασης. Έτσι έχει σταθεροποιηθεί η αγορά και έχει λειτουργήσει πολύ καλά ε, το σύστημα αυτό. Ε, από την εισαγωγή της ρύθμισης αυτής ε, έχουν αναπτυχθεί πολλές οργανώσεις παραγωγών. Συμμετείχαμε στην χρηματοδότηση ΦΕΟΓΑ, όπου δεν υπήρχε ξεχωριστή χρηματοδότηση για την αλληλεία και τις οργανώσεις παραγωγών. Δεν υπήρχε ευφυΐα στην αγορά, το πούμε Δεν υπήρχαν στοιχεία για την αγορά. Ενώ οι παρεμβάσεις αυτές χρειαζόντουσαν πολύ λίγα χρήματα. Ήταν επίσης σαφέ ότι τα πρότυπα τη αγορά και οι πληροφορία, και η πληροφόρηση των καταναλωτών ε, ήταν ελλειπή και χρειαζόντουσαν βελτίωση η χρηματοδότηση ε, ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών ήταν αδύνατη. Όλα αυτά περνούσαν μέσω των κρατών μελών και όταν οι οργανώσει περιγωγών ε, στα κράτη-μέλη θέλανε από κοινού να ε, αναλάβουν πρωτοβουλίε, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση, διότι το κράτο μέλο Α δεν ήθελε να πληρώσει τι δραστηριότητε που θα ελάμβαναν χώρα στο κράτο μέλο Β και αντίστροφα. Ε, βιωσιμότητα και ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών. Η ΕΑΠΟ ΕΕ ε, συμμερίζεται το όραμα της Κομισιόν, δεν θα πρέπει να βιαστούμε όμως. Αν ε, ήταν τα νέα στοιχεία να τεθούν σε ισχύ αμέσω, τότε όλο το σύστημα θα μπλοκαριζόταν. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Προτείνουμε μία προσέγγιση βήμα προ βήμα. Και καθότι υπάρχουν τόσε οργανώσει παραγωγών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθότι διαφέρουν σε μέγεθο και σε δυνατότητες. Ε, ε, ε, η κάθε οργάνωση παραγωγών έχει διαφορετικό σημείο κίνησης και γι' αυτό είναι σημαντικό για τη μετάβαση τα κράτη-μέλη και οι οργανώσεις παραγωγών να συμφωνήσουν πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να μην μπλοκάρουν τη μετάβαση, αλλά να λειτουργήσει ομαλά. Όσον αφορά την αποκέντρωση, αυτή αποτελεί μέρος του βασικού κανονισμού Ε, έχει όμως ε, και άλλες προεκτάσεις, διότι οι οργανώσεις παραγωγών ε, λειτουργούν σε σε, πολλούς, σε πολλά επίπεδα. Ε, είδαμε ότι η, η μεταρρύθμιση της κοινής, της κοινής αλληλευτικής πολιτικής το 2002 οδήγησε στα περιφερειακά συμβούλια, κάτι που λειτουργήσε πολύ καλά. Για το 2012 η πράσινη βίβλος ε, φαίνεται να έχει σημαντικές φιλοδοξίες όσον αφορά την αποκεντροποίηση, αλλά βλέπουμε πολύ λίγα απτά αποτελέσματα στις προτάσεις και υπάρχει ο κίνδυνος να χώρο στην κατάσταση πριν το 2002 με περισσότερες, ε, ε, ε, με περισσότερες εξουσίες στα χέρια των κρατών μελών, κάτι κάτι που ε, θα ε, αποκλείσει κάποιους ε, ενδιαφερομένους. Ενώ το, τα ΡΑΚ, τα Περιφερειακά Συμβούλια, έχουν δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους και στα κράτη-μέλη να, συνεργάζονται. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε αποκέντρωση για να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση. Υπάρχουν δυνατότητες εντός της συνθήκης. Εάν υπάρχει βούληση υπάρχουν και τρόποι. Όπως ε, σας είπα για τις οργανώσεις παραγωγών, ε, δεν υπάρχει ένα μέγεθος που να κάνει για όλους. Εντό τη ΕΑΠΟ έχουμε πολλέ οργανώσει παραγωγών, κάποιε είναι μεγάλε, κάποιε είναι μικρέ και αντιπροσωπεύουμε και διάφορα είδη αλληλεία όπω είδατε από τα σκάφη μα. Υπάρχει διαφορετικό καθεστώ στο κάθε κράτο μέλο. Οι οργανώσει παραγωγών λοιπόν πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται και πρέπει να ε, ανταποκριθούν στι ε, συνθήκες και γι' αυτό θα πρέπει να υπαγορεύεται, ε, δεν θα πρέπει να υπαγορεύεται η ανάπτυξή τους και η εξέλιξή τους, αλλά θα πρέπει να επιτρέπεται, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά την ταχύτητα και τα επίπεδα. Ε, ο, μηχανισμός παρέμβασης, όπως είπε ο κύριος Μαξουίνη, είναι στοιχείο κλειδί. Η ΕΑΠΟ λέει όχι στην ενίσχυση για την καταστροφή τροφίμων, αλλά με το παρόν ε, σύστημα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ε, και ε, στην νέα πρόταση θα συμπεριληφθεί μηχανισμός παρέμβασης για μη ανθρώπινη κατανάλωση. Ο μηχανισμός παρέμβασης αποτελεί ένα πολύ καλό δίκτυο ασφαλείας ε, υπάρχει κίνδυνος όμως για, την αλία μικρής κλίμακες και επί ε, δεκαετίες η παρέμβαση έχει παίξει σημαντικό ρόλο και ε, δεν υπάρχει επιθυμία να καταργηθεί. Μιλάμε για λίγα χρήματα με τεράστια θετικά αποτελέσματα. Και ε, εδώ υπάρχει αντίφαση με την απαγόρευση των απορρίψεων, διότι ε, έτσι καταστρέφονται ψάρια για κανένα σκοπό. Ενώ με, με το μηχανισμό παρέμβαση, ε, η αντιμεταποίηση των ηχθείων για μία ανθρώπινη κατανάλωση, βλέπουμε θετικά αποτελέσματα. Και οι οργανώσει παραγωγών θέλουν να δημιουργήσουν αδεχτή ασφαλεία για τα μέλη του. Και τώρα φτάνουμε σε ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα ε, το στενό μονοπάτι που μας οδηγεί μέσα από τον νόμο του ανταγωνισμού. Οι ε, οργανώσεις παραγωγών πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες αγορά και ε, τα τα προϊόντα που αποκτούμε από τη φύση είναι πολύ συγκεκριμένα και πρέπει να αποφύγουμε την σπατάλη. Και δεν μπορούμε, δεν έχουμε κάποια δεν έχουμε κάποια μέσα να αντιταχθούμε ε, στις ε, δυνάμεις ε, της αγοραστικής δύναμης. Εγώ είμαι Ολλανδός και ξέρω ότι οι αρχές ανταγωνισμού κυνηγάνε τους, τα στελέχη των οργανώσεων παραγωγών. Γι' αυτό χρειάζεται σαφής καθοδήγηση προς όφελος και των αλλιών και των παραγωγών. Και όπως σας είπα πριν, ε, η αλληλεία δεν, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον τομέα τηλεπικοινωνιών. Όσον αφορά τις πράξεις κατοξιδότηση, η παρούσα πρόταση είναι ασαφής και ε, η ανάγνωση του εγγράφου EMFF δεν βοηθάει πάρα πολύ. Θα πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο η πρόταση αυτή. Υπάρχουν αναλυτικοί κανόνες σε διαφορετικές αφορμαστικές πράξεις. Υπάρχει ε, ο κίνδυνος όμως να μην υπάρξει διαβούλευση σε αυτή τη διαδικασία. Εάν είναι ασαφές το βασικό κείμενο και όλα αναβληθούν, τότε μπορούμε να καταλήξουμε να πλημμυριστούμε από νέους καλώνες χωρίς ε, να έχει ε, προηγηθεί η διαβούλευση. Γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη της δέσμευσής μας, διότι ε, πρέπει να βελτιωθεί η ασφάλεια, η βεβαιότητα στον τομέα αυτών. Η ΑΚΦΑ είναι Συμβουλευτική Επιτροπή για, την Αλληλεία. Η ομάδα εργασίας 3 είναι ο μόνος χώρος όπου συναντούνται και συνομιλούν οι αγορές. Εάν λοιπόν διαλυθεί η ΑΚΦΑ, ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιπλέον ε, συμβούλιο αγορά, διότι θα πρέπει οι συμμετέχοντε στην αγορά να μπορούν να ε, συζητάνε την κατάσταση μεταξύ του. Και θα πρέπει αυτό να υπάρξει πριν την κατάργηση τη ΑΚΦΑ, διότι αλλιώ θα δημιουργηθεί κενό. Η ΕΑΠΟ θα υποβάλει αναλυτική πρόταση μαζί με τους εταίρους μας στην αγορά και κάτι τέτοιο θα συμπεριλάβει και προτάσεις για την ε, σύσταση και τους σχετικούς κανόνες. Όσον αφορά τις ε, απορρίψεις, ε, αυτό υπόθηκε και πριν. Οι οργανώσεις παραγωγών έχουν τώρα ένα νέο καθήκον, το οποίο όμως δεν τους αρέσει καθόλου. Θα πρέπει να ασχοληθούν με τα αναπιθύμετα αλλιεύματα, θα πρέπει να εφαρμόσουν κανόνες για την εξάλληψη των απορρίψεων ε, μιλάμε για τεράστιες οικονομικές ε, συνέπειες και το ξέρω αυτό από τις κάτω χώρες όπου ε, το κόστος για τον τομέα είναι 10 με 18 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι πολύ καλή προσέγγιση διότι έχουμε θνησιμότητα των ηχθείων κατά 100%. Χρειάζεται λοιπόν να απαγορευτούν οι απορρίψεις. Σημαντικό είναι ε, η αποφυγή, η ελαχιστοποίηση και τα κίνητρα. Όσον αφορά το EMFF και τη χρηματοδότηση, ε, πολύ μεγάλο μέρος της διαδικασίας, ε, να πω και στα κράτη-μέλη, απαιτείται προσανατολισμός, όχι υπαγόρευση, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο προσανατολισμό. Η οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει λόγο για τα κράτη-μέλη να μην ε, συγχρηματοδοτήσουν. Εάν λοιπόν οι οργανώσεις παραγωγών ε, ε, επιλέξουν την συγχρηματοδότηση, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ιδιωτική συγχρηματοδότηση. Όσον αφορά τις μεταβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις, κάποια μέλη της ΕΑΠΟ ε, ε, βρίσκονται στον πυρήνα ε, της συνδιαχείρισης. Από μόνες τους οι παραχωρήσεις αυτές δεν θα λειτουργήσουν. Έχουμε το παράδειγμα της Δανίας και των κάτω χωρών που δείχνουν ότι μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέτρα θα αποτελέσουν επιτυχία οι μεταβιβάσιμες παραχωρήσεις. Στις χώρες αυτές πράγματι έχουν αποτελέσει σημαντική επιτυχία. Αυτό το έχει παραβλέψει το ελεγκτικό συνέδριο να ε, προβλέπονται οι παραχωρήσεις αποκλειστικά για ενεργούς αλληλείς ε, και κλείνοντας Είμαστε υπέρ ε, νέας ρύθμισης, διότι η παρούσα δεν ε, ε, ε, ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Η ΕΑΠΟ θέλει νέα, νέο κανονισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις μερωτικές εξελίξεις και η ΕΑΠΟ προσφέρει μια πλατφόρμα για ανταλλαγή των απόψεων υπό το φως αυτών των εξελίξεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βίσερ και θα δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Πολινάριο που είναι ο τελευταίος ομιλητής ε, για αυτό το σκέλος. Για αυτό το πάνελ έχετε το λόγο. Ici, après sur un Oh, micro. Um, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν ε, να, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία που αναλάβατε ως Επιτροπή Αλίας, αλλά επίσης θα ήθελα να απευθυνθώ και στην κυρία Φράγα που είναι παρούσα εδώ, είναι, είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό και θέλω να τη στείλω ένα χαιρετισμό. Και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Πατράου Νέβες ε, που μου ζήτησε να παρευρεθώ εδώ και τον κύριο άντες ε, που είναι συνταξιδιώτης μου για πάνω από 20 χρόνια. Και θα ήθελα να πω το εξή ε, Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο βάσει του θέματος που μου προτείνεται. Είμαι ε, εκπρόσωπος της Πορτογαλικής προσωπίες ε, της ε, Πορτογαλικής Διεύθυνσης ε, Αλίας, όμως δεν σημαίνει το ότι τόσο θα πω είναι πολιτικά. Επίσης, μετά τις δύο παρεμβάσεις που ακούστηκαν εδώ, θα ήθελα να πω ότι θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε τρεις άξονες. Στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών, την βελτίωση της παροχής των πληροφοριών στους καταναλωτές και στην, στο να δοθεί μεγαλύτερη ε, αξία, να δειχτούν περισσότερα τα ελευτικά προϊόντα. Όπως όλοι γνωρίζετε... Ε, Μάλλον όλοι γνωρίζετε από πού προερχόμαστε και σε ποιο πλαίσιο κινείται ο ελευτικό τομέα και καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε τώρα για την κοινή οργανώση αγορά και για τα ελευτικά προϊόντα. Υπάρχει ένα τεράστιο βάρος από τις ε, εισαγωγές ε, και επίσης ε, υπάρχει μεγάλη ετερογένεια των διάφορων ειδών Επίσης, στην οργάνωση αγοράς και στις συνήθειες κατανάλωσης στο σημείο αυτό και πάλι βρισκόμαστε στο γενικό πλαίσιο. Θα ήθελα επίσης να παρουσιάσω δύο σημεία. Ότι υπάρχει μια τάση και αύξηση τη κατανάλωσης των ελευτικών προϊόντων και των ε, ψαριών και φυσικά αυτό σχετίζεται και με θέματα υγεία, η κυρία Επίτροπος ε, υπογράμμισε σε μια διάσκεψη ε, το θέμα των ωμέγα 3 και του βάρου. Η δατοκαλλιέργεια δεν ε, σημειώνει την ανάπτυξη που θα μπορούσε να έχει. Αυτό έχει να κάνει βέβαια όχι με την αγορά αλλά με τη χρηματοδότηση γιατί οι επιχειρήσεις ε, για να λάβουν κοινοτική χρηματική στήριξη πρέπει να είναι μικρέ και μεσές επιχειρήσει. Και κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι αυτή η ε, πτυχή ότι ε, τα προϊόντα αυτά τείνουν να σπανίζουν και κατόπιν έχουμε κάποια στοιχεία της Eurostat από το 2007 και θα ήθελα επίσης να τα παρουσιάσω γιατί εδώ βλέπετε μία προοπτική των δαπανών των ε, οικογενειών ε, στα τρόφιμα. Και εγώ πιστεύω ότι τα αλληλευτικά προϊόντα Ε, καταλαμβάνουν μια μεγάλη θέση στην κατανάλωση. Βέβαια στην πρώτη θέση βρίσκονται Πορτογαλία και Ισπανία, κατόπιν ακολουθεί η Γαλλία και ε, μιλάμε για το 15% παραδείγματο χάρη κατανάλωση σε αλευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Πορτογαλία παραδείγματο χάρη φτάνουμε στο 49%. Σε ό,τι αφορά τι οργανώσει παραγωγών, εγώ πιστεύω ότι η γενική στόχη τη πρόταση ε, για την ΚΟΑ σήμερα μπορούμε να ε, τις υποστηρίξουμε. Όμως υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ε, έναντι των προκλήσεων που θέτει η αγορά. Καταρχήν, πρέπει να εγγυθούμε μεγαλύτερη απλούστευση και διασύνδεση με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής ε, και επίσης πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε επικαλύψεις ενιών που οδηγούσαν σε σύγχυση και σε αυξημένο δικαιωτικό κόστος της εφαρμογής. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για να έχουμε μία μεταρρύθμιση της ΚΟΑ και ταυτόχρονα Ε, να επιτρέψουμε να λειτουργεί αυτό χωρίς ε, βέβαια ε, να έχει καθοριστεί το κονδύλι και αυτό είναι μια επιφύλαξη που θέλω να καταθέσω εγώ εδώ. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τα μέτρα αγοράς, υπογραμμίζω την απόλυτη απουσία οποιασδήποτε προσέγγιση σε θεμάτων του, του εξωτερικού κεφαλαίου, της εξωτερικής πτυχής. Η Κομισιόν λέει ότι υπάρχει διαφορετική νομική βάση, όμως εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι στην πρόταση που έχουμε επιτάπητος ε, λείπει πλήρως αυτή η αναφορά στην εξωτερική πτυχή και νομίζω ότι εδώ πρέπει να κινηθούμε προσεκτικοί γιατί έχουμε πολλές εισαγωγέ Για το παρατηρητήριο της αγοράς που παρουσιάζεται ως μια λύση για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό πρέπει να το προωθήσουμε, να το πληστοποιήσουμε, πρέπει να διαδίδουμε καλύτερα τα στατιστικά δεδομένα, όμως δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε προς μια βαριά δομή η οποία ε, θα επικαλύπτεται με άλλες. Ε, και σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, ε, καλό θα ήταν να υπάρχει μια κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ του θεσμικού ρόλου των διάφορων οργάνων και πρέπει να έχουμε περισσότερη συναπόφαση και λιγότερες κατεξουσιοδότηση πράξης. Άλλο σημείο που θα ήθελα να φέρω ε, είναι οι νέες προκλήσεις που τίθενται. Καταρχήν, να υπογραμμίσω ότι παρά το ότι υπάρχουν παγιωμένε οργανώσει παραγωγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει εμείς από τεχνική και οικονομική σκοπιά να παγιώσουμε το ρόλο αυτών των ε, οργανώσεων παραγωγών. Ε, η αναγνώρισή τους θα πρέπει ε, να προκύπτει από τον αριθμό των μελών ή από τις δραστηριότητές τους. Δεν μπορούμε απλώς να μιλάμε για μείωση των οργανώσεων παραγωγών γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στο να μειωθούν τα μέλη όταν πρέπει να ακολουθήσουμε εντελώ διαφορετική οδό. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν οι προποθέσει για να υπάρχουν περισσότεροι αλλοί στην αλία μικρή κλίμακα. Και επίση μα φαίνεται σημαντικό να χαιρετήσουμε ε, το, την δυνατότητα να παρουσιάζονται τέτοια σχέδια διαχείρισης και από τις κοινοπραξίες οργανώσεων παραγωγών. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι μία οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε, πρέπει να τη χαιρετήσουμε και θα ενισχύσει το ρόλο των οργανώσεων παραγωγών. Σε ό,τι αφορά ε, τώρα τις απορρίψεις, αν ε, λάβουμε υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει κάτι που άλλε χώρε η Νορβηγία λόγου χάρη, χρειάστηκε 20 χρόνια για να ελοποιήσει και που εμεί προτείνουμε τώρα να το κάνουμε σε 2-3 χρόνια, εδώ πράγματι υπάρχει ένα θέμα κλειδί. Δηλαδή να δημιουργηθούν οι προποθέσει έτσι ώστε οι οργανώσει παραγωγών να μπορούν να έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο ή να μπορούν να συμμετέχουν στην επίτευξη αυτού του καθολικού στόχου τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛΠ. Και τώρα μου φαίνεται υπερβολική αυτή η οριζόντια θέση ε, που έχει ληφθεί. Και γι' αυτό ακριβώ θέλω να επισημάνω κάτι που μου φαίνεται παράλογο και είναι το εξή. Σήμερα, μέσω ενός ε, μηχανισμού αποσύρσεων, ή οργανώσει παραγωγών μπορούν να προχωρήσουν ε, στο να χορηγούνται, να δίνονται αυτά τα ελευτικά προϊόντα σε φιλαστροφτικές οργανώσεις. Αν δούμε την πρόταση κανονισμού που έχει κατατεθεί, ε, σε τι μας οδηγεί, ότι ε, αυτά τα ψάρια τα οποία ε, τελικά είναι μικρότερου μεγέθους ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει τελικά να καταστρέφονται, να χρησιμοποιούνται και χθέλευρα και δεν μπορούν να δίνονται πλέον στις οργανώσεις γιατί για να μην δημιουργηθεί μια παράλληλη αγορά όμως ε, σήμερα πρέπει να προσέξουμε ότι οι οργανώσεις παραγωγούν παραγωγών ε, χρησιμοποιούν αυτό το μηχανισμό απόσυρση για να προσφέρουν τα προϊόντα σε φιλανθρωπικέ οργανώσει. Και αυτό λαμβάνει χώρα σε στιγμέ ύφεση, όπω ζούμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τελευταίο σημείο. Οι οργανώσει παραγωγών πρέπει επίση να μπορούν να προωθήσουν την παραγωγή του. Και αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για την ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών. Τώρα, αν στραφούμε στο πώς ε, θα δώσουμε μεγαλύτερη αξία στα λευτικά προϊόντα, πώς θα αναδείξουμε περισσότερο τα προϊόντα αυτά. Εμείς ε, ξεκινάμε με την προϋπόθεση ότι εδώ έχουμε τέσσερις θεμελιώδεις άξονες. Δηλαδή ότι προέρχονται τα προϊόντα αυτά από ένα φυσικό περιβάλλον, τα ψάρια προέρχονται από ένα φυσικό περιβάλλον και εμείς ε, πρέπει να υπερασπίσουμε αυτή τη σκοπιά δηλαδή πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκό το ε, το καλλιέργεια και αλίας. Πολλές φορές ε, στην αγορά, η αγορά μας κατακλείζεται από προϊόντα που παρουσιάζεται ε, όπως, από ψάρια όπως είναι ο παγκάσιο ή η υπέρκα του Νείλου Όμως ε, εδώ θεωρώ ότι εμεί πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς να αναδείξουμε τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη ερώτηση, δηλαδή, έχουμε πρώτο θέμα, έχουμε ε, την προπόθεση ότι προέρχονται από ένα φυσικό περιβάλλον τα ψάρια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία του είδους ε, για την τοπικό πολιτισμό και την κουζίνα, την τοθεσία, Πρέπει να έχουμε πιστοποίηση των προϊόντων και περισσότερες λεπτομέρειες στις ετικέτες και πρέπει να χρησιμοποιούμε τις καλές ε, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές. Λοιπόν, ε, τώρα όταν λέμε προέλευση, γιατί δεν βάζουμε τη χώρα ή το λιμάνι εκφόρτωσης, παραδείγματος χάρη, Οι φυστάμενε λύσεις ε, είναι εξή. Κάθε κράτο μέλος ε, προσπαθεί ε, να βρει τρόπους για να αναδείξει περισσότερο τα αλληλευτικά προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για τι ενώσει παραγωγών. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι μέχρι πού πρέπει να φτάνουμε στις πληροφορίες που παρέχουμε. Εγώ θεωρώ ότι ε, θα πρέπει οι πληροφορίες ε, να καλύπτουν τα πάντα. Δηλαδή, από τη ε, στιγμή της αλίευσης μέχρι το πιάτο. Πρέπει να έχουμε και υπεύθυνη κατανάλωση. Έτσι, λοιπόν... Αν υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος όταν αυτό πωλείται, όταν εκφορτώνονται, ε, και στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε αυτές τις πληροφορίες ακόμη και στο εστιατόριο γιατί μπορεί ο καταναλωτής να έχει πλήρες πληροφορίες για το τι καταναλώνει, για το τι τρώει. Και επίσης είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, να δούμε ε, το θέμα της υποχρεωτικής ετικετοθεσίας και της εκούσιας ετικετοθεσίας. Η πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ ξεκαθαρίζει ε, τι πρέπει να καλύπτεται από την ε, υποχρεωτική ετικετοθεσία και μετά υπάρχει και ένα τμήμα για την εκούσια ετικετοθεσία. Τώρα για την εκούσια ετικετοθεσία ε, είναι η ετικετοθεσία των κατευθύνων γραμμών της ΦΑ. Ορισμένα θέματα είναι πιο λεπτομερή και πιο συγκεκριμένα από όσα προβλέπονται στην υποχρεωτική ε, ετικετοσία. Πρόκειται για τοσία που έχουμε ε, δυνάμει παραδείγματο χάρη του Συμβουλίου Επιστασία της Θάλασσα, ε, το MSC. Σε περιπτώσεις αυτές έχουμε περισσότερες απαιτήσει από αυτά που προβλέπονται στην υποχρεωτική νομοθεσία. Λοιπόν, η εκούσια ετικετοσία θα πρέπει να θέσει κάποια ελάχιστα πρότυπα Και βέβαια εδώ ε, ίσως ε, θα έπρεπε να παρέχουμε και περισσότερες διατροφικές πληροφορίες, ε, δηλαδή πώς ε, τα ψάρια ωφελούν την υγεία και να συνδέσουμε έτσι το θέμα της διατροφής με την υγεία. Και τέλος δεν μας φαίνεται καθόλου απαραίτητο να υπάρχει επιβολή νέων ε, κανόνων, νέων προτύπων αντικαθεσία για ε, τις κονσέρβες, παραδείγματο χάρη, κονσέρβες τόνου ή Σαρδέλε. γιατί εκεί υπάρχει ήδη συγκεκριμένη ρύθμιση που έχουμε στον κανονισμό του 89 και του 2002. Και τέλος, για να ολοκληρώσω, θα έλεγα ότι η ανάδειξη των ελευτικών προϊόντων, των προϊόντων ελίας και η ευθυγράμμιση με τη στρατηγική για το 2020 έγκυται ε, σε αυτές τις δηλαδή να αποδείξουμε την ποιότητα, περιβαλλοντική ευθύνη, βιωσιμότητα της ελίας και σύνδεση της κατανάλωσης ψαριού με την καλή υγεία. Αλλά επίσης να αυξηθεί και η διασύνδεση των οργανώσεων παραγωγών με τη διανομή και να ενισχυθεί ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την τοπική και την ερασιτεχνική αλία. Και επίσης ε, διάρθρωση μεταξύ της παράδοσης και της ε, ζήτησης ε, και αυτό από την πλευρά των πιο νέων, γιατί εδώ πρέπει και να καταπολεμήσουμε ε, μάλλον πρέπει να οθήσουμε τους νέους να καταναλώνουν ε, προϊόντα ελίας και επίσης γνωρίζετε ότι έχουμε και προβλήματα δημόσιας υγείας, έχουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας και ε, δυστυχώς αυτά τα προβλήματα ξεκινούν πλέον ε, στους πιο νέους. Επίσης, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση για την τιμή του προϊόντος, κυρίως από την πρώτη πώληση, την, τιμή πρώτης πώλησης, Μάλιστα, το παρατηρητήριο είπε ότι αυτή η αρχή είναι ιδιαίτερα σωστή, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες ε, για την τιμή πρώτης πώληση, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε ε, την απόδοση και το εισόδημα των αλλιέων. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πολυνάριο. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι παρεμβάσεις των τριών ε, πρώτων προσκεκλημένων και θα ξεκινήσουμε ένα γύρο παρεμβάσεων ε, για τους βουλευτές που επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Ποιος θα ήθελε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι διαφαίνεται σιγά σιγά μία συνένεση για την δυνατότητα να συνεχίσουμε με το μηχανισμό τιμών παρέμβασης σύστημα στο οποίο έχει επιτεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι θέλει να έχει έναν ενιαίο μηχανισμό αποθεματοποίησης, αποθήκευσης, που χρησιμοποιείται σε κάποια νότια κράτη-μέλη και όχι τόσο πολύ στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντί να υπάρχουν ελάχιστες τιμές και σχετικές ε, ε, μέτρα παρέμβασης θα υπάρχουν κάποιες τιμές εκκίνησης κάτω των οποίων ορισμένα είδη θα καταψύχονται και θα αποθηκεύονται. Ως προς την πρόταση αυτή, είδα ότι υπάρχουν αρκετά αμφιλεγόμενες αντιδράσεις. Υπάρχουν πολλοί που στηρίζουν ε, τη συνέχιση του συστήματος του μηχανισμού των τιμών. Άλλοι λένε ότι αυτό οδηγεί σε υπεραλίευση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει ενδεχομένω ο κύριος ε, Μαξουίν και ο κύριος Βίσερ ποια είναι η δική τους η άποψη όσον αφορά το σύστημα αυτό του trigger price των τιμών εκκίνησης καθώς επίσης και του ενιαίου μηχανισμού αποθήκευσης που περιλαμβάνει και ένα τμήμα κατάψυξης. Αναφερθήκαν και οι δύο στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς όμως να αναφερθούν συγκεκριμένα στο μηχανισμό τιμών εκκίνησης. Νομίζω ότι καλύτερα να ακούσουμε πρώτα όλες των βουλευτών και στη συνέχεια να δώσουν τις απαντήσεις ε, ομαδοποιημένα οι ομιλητές, γιατί φαντάζομαι ότι θα συμπίπτουν κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Φράγα. Εγώ από τις περιβάσεις ε, κυρίως των δύο πρώτων ομιλητών, ε, μπορώ να σας πω ότι μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι αυτοί αναφέρθηκαν ε, κυρίως στο θέμα των απορρίψεων και τι θα σημαίνει για αυτούς ε, να ασχοληθούν με, ακριβώς με αυτό το θέμα που τίθεται τώρα στην ΚΟΑ. Και οι δύο μιλητές που αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό είπαν ότι είναι κατά της απαγόρευσης των απορρίψεων. Και ότι θα ήταν ε, υπέρ του να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις απορρίψεις. Αυτό θέτει σημαντικά προβλήματα γιατί το οικονομικό ζήτημα, δηλαδή το κόστος ε, που μπορεί να υποθέτει όλο αυτό για τις οργανώσεις παραγωγών, νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται στο νέο χρηματοοικονομικό κανονισμό, αν και δεν είναι πολύ σαφές Απλώς κατά κάποιο τρόπο λέγεται ότι θα υπάρχει χρηματοδότηση. Όμως ούτε καν ξέρουμε μέχρι ποιο ποσό και με ποιο τρόπο. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν να καλυφθεί από το χρηματοοικονομικό κανονισμό. Αλλά αν ε, για σας η διαχείριση των απορρίψεων αποτελεί ένα ανεπίλητο πρόβλημα, τότε εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Για το θέμα των παρεμβάσεων. Θα ήθελα να μου πείτε αν ε, όλοι οι μηχανισμοί παρέμβαση θα μπορούσαν να μειωθούν περισσότερο. Εγώ θα συμφωνούσα εδώ περισσότερο με την πρόταση τη Κομισιόν, για να είμαι ειλικρινή. Αν από την πλευρά των οργανώσεων παραγωγών υπήρχε μεγαλύτερος σχεδιασμός ε, της παραγωγής. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τώρα τα επιχειρησιακά σχέδια δεν μπόρεσαν να προετοιμαστούν καταλήλως από τις οργανώσεις παραγωγών, έλλειψη επιλεξικότητας, ε, ε, έλλειψη πρόβλεψης, τη ζήτηση της αγοράς, καλύτερη διαχείριση θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μία λύση. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν οι οργανώσει παραγωγών ε, μπορούν και είναι σε θέση να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα έπρεπε να προετοιμάσουν αυτά τα σχέδια με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Όμω νομίζω ότι οι περισσότερε ε, τέτοιε μικρέ οργανώσει παραγωγών δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Ήθελα να το αναφέρω και αυτό, αλλά αυτό που με ανησυχεί κυρίω είναι το θέμα των απορρίψεων. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω πολύ καλά πώ ε, θα ολοκληρωθεί αυτό, αλλά φυσικά ο τομέα, ε, ο κλάδο είναι ο πρώτο που γνωρίζει πώ μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα τη απαγόρευση των απορρίψεων. Και αυτή η απομάκρυνση τη ε, δική σα θέση από τη θέση της Κομισιόν ε, είναι κάτι που μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό και μου προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Ευχαριστούμε κυρία Φράγκα. Κύριε Γκάλαγκερ. Ε, ε, Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, όλους τους ομιλητές. είναι προφανές ότι έχουν άμεση πείρα με τα θέματα αυτά. Η ε, οργανώσεις παραγωγών ε, επί σειρά ετών έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ε, κατά την διατήρηση των επιπέδων των τιμών. Έτσι μπόρεσαν να επιβιώσουν και η αλληλεία και οι αλληλείς. Γιατί όμως ήταν τόσο απαραίτητες, ιδιαίτερα στον πελαγικό τομέα, επειδή δεν υπήρχε πραγματική ρύθμιση όσον αφορά τα αλλιεύματα και τις εκφορτώσεις. Δεν υπήρχε προσπάθεια να ε, ε, είναι αναλογική η ε, ικανότητα στη, σε αυτές με τις εκφορτώσεις και σε περίπτωση που είχαμε ταυτόχρονες εκφορτώσεις πολλών ηχθείων ε, έπρεπε πολλά από αυτά να χρησιμοποιηθούν για τα αλευρά. Θα πρέπει να μάθουμε όμως από τις εμπειρίες μας και να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στις οργανώσεις παραγωγών. Ξέρω από τη δική μου χώρα ότι παρεμβαίνουν και προσπαθούν να πείσουν τα σκάφη να μην φτάνουν όλα ταυτόχρονα ανάλογα με την ε, ικανότητά τους ε, και τη ζήτηση. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο τομέας της αλληλείας θα επικροτήσει κάτι τέτοιο. Ίσως θα μπορούσε μια τέτοια πρόταση να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ε, δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαι εδώ, άλλο θα είναι περισσότερο, άλλο θα είναι λιγότερο, αλλά μιλάμε πάντα για τα αλλιεύματα. Το θέμα είναι η τεχνική συντήρηση των ε, ε, αποθεμάτων, διότι όπως είπα το πρωί στην πρόεδρο του Συμβουλίου, ε, ο μόνος τρόπος να μειώσουμε τελείως, να εξαλείψουμε τελείως τις απορρίψεις είναι να σταματήσουμε να ψαρεύουμε. Αυτό βέβαια είναι υπερβολικό. Ε, εγώ είμαι αποφασισμένος να αγωνιστώ για την ε, μείωση και την εκφόρτωση ε, των απορρίψεων. Αλλά εάν υπάρχει απαγόρευση για κάποιο είδους ε, ε, ηχθείων ε, εάν αλλιευτούν δεν υπάρχει κάποια λύση. Αυτό που ουσιαστικά λέμε θα πρέπει να εκφορτωθούν δηλαδή. Όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις αγορές, αλλά Πολλοί από τους φορείς για τους οποίους μιλάμε ε, μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην αγορά και έχετε δίκιο ότι η 100% δεν βοηθάει κανέναν. Προσπαθώ λοιπόν να πω πρώτον να σκεφτούμε μήπως πρέπει να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στις οργανώσεις παραγωγών ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στις ρυθμίσεις υπάρχει μια άτυπη ε, ρύθμιση η οποία όμως δεν ε, βοηθάει. Ε, στην Ιρλανδία και στη Σκοτία στις 2 Ιανουαρίου. Αλλιεύουν όλα τα σκάφη, όλα φτάνουν ταυτόχρονα και οι εκφορτώσεις ξεπερνάνε κατά πολύ την ε, δυνατότητα μεταποίησής τους. Ας μάθουμε τουλάχιστον αυτό, να ρυθμίζουμε δηλαδή τα αλλιεύματα και τις εκφορτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήτανε πολύ καλές οι ομιλίες. Εάν θα μπορούσε η Γραμματεία παρακαλούμε να μοιράσει τις ομιλίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ε, αφομοιώσουμε όλα τα στοιχεία αυτά στο τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Σφεραίρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα και το πρωί και χθες και εγώ θεωρώ ότι αυτή η ακρόαση και αυτές τις ε, τρεις παρεμβάσεις που ακούσαμε Αναμφισβήτητα και οι τρεις εμπλουτίζουν τη συζήτησή μας. Εγώ ήθελα απλά να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τόσο αναφέρθηκαν εμείς. Ε, είχαμε την ευκαιρία, όπως σας είπα, να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με μακρόν και θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με μία από τις τυχές ε, που αναφέρθηκαν από όλους τους ομιλητές με το θέμα ε, των εσόδων. Ε, κάποιος είπε ότι δεν θα υπάρχει βιώσιμη αλία αν δεν είναι και το εισόδημα αξιοπρεπές ε, για τους αλείς. Και αυτό είναι ένας γορδίος δεσμός που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας, ο κλάδος και αν δεν το λύσουμε αυτό το θέμα δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε και άλλα ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το τι γίνεται ε, με τις ε, αποσύρσεις ε, και ένας από τους στόχους της αλληλευτικής πολιτικής ήταν να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα οι γεωργοί, όμως απέτυχε η κοινή αλληλευτική πολιτική. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια μεταρρύθμιση η οποία τελικά να μπορέσει να πετύχει τους στόχους που δεν έχουν καλυφθεί και η πρόταση της Κομισιόν που έχουμε σου ούτε αυτή μας δίνει μια ικανοποιητική απάντηση για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε αυτή την πτυχή. Και Επίσης, ε, ο εισηγητής πάντα θέτει το θέμα ε, που αφορά την οικολογική ετικέτα και πώς μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες πληροφορίες στον καταναλωτή για να δείξουμε το τελικό προϊόν. Και ο κύριος από την Πορτογαλία ανέφερε το θέμα της ε, ονομασίας προέλευσης και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ε, να το φροντίσουμε αυτό και να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη σκέψη λοιπόν ήθελα να κάνω εδώ. Είναι σπάνιο είδος ε, το ψάρι και βλέπουμε ότι αυξάνεται η αξία του, αναδεικνύεται το λένε και περισσότερο για διάφορους λόγους και τελικά εμείς μας ενδιαφέρει να προσδώσουμε αξία στο τελικό προϊόν. Όμως έχουμε πάρα πολύ χαμηλές τιμές στην πρώτη πώληση και αυτό είναι αλήθεια και ο τελικός καταναλωτής πληρώνει ακριβά. έτσι λοιπόν ε, <laughs> μπορείτε να βάλετε όποια ετικέτα θέλετε, οικολογική ή όχι, η τιμή είναι αυτό που καθορίζει αν θα το αγοράσει ο καταναλωτή. Έχουμε λοιπόν ενισορροπία, προφανή ενισορροπία στην αλυσίδα, χαμηλέ τιμέ στην πρώτη πώληση και υψηλέ τιμέ στον τελικό καταναλωτή γενικά. Υπάρχουν διάφορες στρεβλώσεις που εισάγονται, ε, έχουμε και τις εισαγωγές και Επίσης, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παρεύουμε σε αυτή την αλυσίδα έτσι ώστε να επιτρέψουμε καλύτερη και πιο δίκαιη κατανομή ε, της αξίας όλη την αλυσίδα. Γιατί το θέμα που τίθεται πάντα είναι ε, τα μέγιστα περιθώρια ε, της θέσης εμπορίας. Υπάρχουν διαφορές, πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση ε, με τη θέση σε εμπορία, τις δομές σε εμπορίας, όμως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν ε, πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια στους ενδιάμεσους. Και υπάρχει ένας ε, τρόπος να το διορθώσουμε αυτό και να θέσουμε κάποια ανώτατα όρια εμπορίας και αυτό θα εγγυθεί μια εξέλιξη. Διάφορα κράτη-μέλη όπως η Πορτογαλία έχουν σχετική εμπειρία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και μεγαλύτερη τιμή πρώτης πώληση, θα έχουμε συγκράτηση της τιμής στον τελικό καταναλωτή. Έτσι λοιπόν θα κερδίσουν ε, τα δύο κράτη αλυσίδας ε, περισσότερο. και θα υπάρχουν και καλύτερη κατανομή στο σύνολο της αλυσίδα. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές. Άκουσα πολλά από τους ομιλητές όσον αφορά τις τιμές παρέμβασης ότι είναι απαραίτητες προκειμένου να πετύχουμε μια κάποια σταθεροποίηση, ιδίως όσον αφορά τους μικρούς στόλους που εξαρτώνται πάρα πολύ από αυτές τις τιμές και το καθεξής. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει, τι θα μπορούσε να συμβεί με τις τιμές παρέμβασης. ένα παράδειγμα του πόσο άσχημα λειτουργεί η αγορά και του πόσο θα μπορούσε τελικά να βελτιωθεί ακόμα και ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών. Θα αναφερθώ στο παράδειγμα της γλώσσας στη Δανία. Η γλώσσα είναι ένα είδος αντικείμενο υπεραλίευσης τα τελευταία χρόνια. Έχει εξαντληθεί σχεδόν το απόθεμα γλώσσας. Και αφού πέρασαν κάποια χρόνια καλής ανασύστασης του αποθέματος αυτού, ξαφνικά εγκαταλείφθηκε το είδος το 2010, μάλλον το 2010 ξαφνικά η Δανία ε, αλίευσε 7.500 τόνους γλώσσας, εκ των οποίων 1.832 πήγανε για καταστροφή που πλήρωσαν τελικά οι Ευρωπαίοι φορολογόμενοι. χρησιμοποιήθηκε μια κίτρινη μπογιά πάνω στο είδος αυτό. Δεν προορίστηκε προς την δετοκαλλιέργεια και 1832 τόνοι γλώσσες αστικά καταστράφηκαν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο δανέζικος στόλος στράφηκε κατά, μάλλον, μάλλον της γλώσσας αυτής, μολονότι δεν υπήρχε αγορά συγκεκριμένη για τη Δανία. Στη Γερμανία 17 ήταν οι αντίστοιχοι τόνοι. Επομένως, οι 1832 θα μπορούσαν ουσιαστικά να είχαν διοχετευθεί στη Σουηδία, στη Γερμανία, σε κάποια γειτονική χώρα και κάπου αλλού. Αλλά είδαμε ότι μια λύση αντιμετώπισε ουσιαστικά ένα διαρθρωτικό πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες επιδοτήσεις ε, για τα καύσιμα, υπάρχουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις εξαιτία της κακοκαιρίας. Όλα αυτά όμω συναθρίζονται και τελικά ενδεχομένω να είναι οικονομικά συμφέρον για τους αλείς να αλλιεύουν ήδη μόνο και μόνο για την τιμή παρέμβασης. Αυτό είναι απαράδεκτο, ιδίως απέναντι στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Μα εξοργίζει λοιπόν η κατάσταση αυτή και ήδη οι πολίτε τη Δανία έχουν εξοργιστεί με την κατάσταση αυτή. Το ίδιο έχει συμβεί με τι Γαρίδε στην Σουηδία, έχει συμβεί με τον Γάδο επίση στη Σουηδία και σίγουρα τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να επαναληφθούν στο μέλλον. Η πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να έχουμε κάποιου μηχανισμού αποθήκευση, την πρόταση αυτή μπορούμε να την αποδεχθούμε, αλλά και οι αλληλεί από τη δική του την πλευρά θα πρέπει να κάνουν κάποιον σχεδιασμό, ένα κάποιο προγραμματισμό και να αλλιεύουν με βάση τι ανάγκε τη αγορά. Διαφορετικά, μην αλλιεύουν. Διαφορετικά, καταλήγουμε εμεί να επιδοτούμε κάποιε ε, άχρηστες αλλιευτικέ δραστηριότητε ή την αλλίευση ειδών που δεν χρειάζεται τελικά η αγορά. Ευχαριστούμε, κύριε Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα αναφερθώ σε κάποιες πτυχές, μάλλον χωρίς να αναφέρω πτυχές που αναφέρουν οι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω δύο τινά. Το πρώτο, έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών. Αναφέρθηκε αυτό εδώ και υπόθηκε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε περισσότερε εξουσίε, αρμοδιότητε ε, στι οργανώσει παραγωγών, αλλά και να δούμε ποιο είναι ο ρόλο του. Και εδώ θα συμφωνούσα 100% με την κυρία Φράγκα που είπε ότι ήταν σημαντικό, ότι είναι σημαντικό οι οργανώσεις παραγωγών ε, να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο σχεδιασμό. Θα ήθελα βέβαια να κάνω ένα βήμα παραπέρα και να μιλήσω για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Γιατί βλέπουμε τελικά ότι δεν ε, είναι μόνο απαραίτητο σχεδιασμό σε επίπεδο παραγωγής, αλλά ε, σε όλο τον τομέα, σε όλο το για να καλύψουμε όλο τον τομέα, παραδείγματο χάρη, η βιομηχανία τη κορσοφοβία πολλέ φορέ χρειάζεται ψάρια και δεν έχει γιατί δεν υπάρχει ε, προμήθεια. Δεν υπάρχουν προμηθευτέ για διάφορου λόγου που του γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι πρέπει να επενδύσουμε όχι μόνο ε, στο να δώσουμε περισσότερες εξουσίε στι οργανώσει παραγωγών και να απαιτούμε μεγαλύτερη παρέμβαση από αυτές σε επίπεδο ε, σχεδιασμού, αλλά να προχωρήσουμε και για τις διεπαγγελματικέ οργανώσει. Καμία καινοτομία δεν αποτελεί αυτό, γιατί τελικά είναι μια διαδρομή που ήδη ακολουθούνται στη ε, γεωργικό τομέα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στις κοινοτικές πολιτικές έχουμε παράλληλες προσπάθειες που γίνονται σε διάφορους τομείς. Κάτι άλλο τώρα στο οποίο θέλω να επισημάνω. Έχει να κάνει με τον προορισμό των ε, των αλλιευμάτων, ε, γιατί άκουσα νομίζω εδώ αντικρούμενες απόψεις ε, μεταξύ των ειδικών αφενός. Εγώ Κατάλαβα ότι αναφέρθηκε κάποιο στη δυνατότητα να παρέχονται σε φιλανθρωπικές ε, οργανώσεις ε, αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να οδηγήσει σε τρέβλε αγοράς, όμως κάποιος άλλος υποστήριξε ότι αυτή θα ήταν μια πιθανή οδός. Αυτό που φαίνεται με ένα ουσιαστικό και που υπόθηκε για την κυρία Φράγα είναι το εξής υποτίθεται ότι ο τομέας ε, πρέπει να έχει ε, μια καθαρή εικόνα αυτού του προβλήματος, δηλαδή των περιπτών ελευμάτων. Ε, δεύτερον, να θέλει να παρέμβει με ένα αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να εξαλειφθούν όσο το δυνατό περισσότερο ε, τα παραλιεύματα. Όπως είπε ο κ. Κάλλανκερ, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να έχουμε μηδενικά απαρρίπτονται αλλιεύματα, τουλάχιστον εκεί όπου έχουμε πολλαπλά είδη όπου αλλιεύονται και επίσης ε, να βρεθούν και να εφαρμοστούν κάποιες λύσεις να συνεισφέρει και ο κλάδος έτσι, όλοι μας, έτσι ώστε όλοι μας από κοινού να μπορούμε να καταθέσουμε προτάσεις που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματική μείωση των περιπτώτων ελευμάτων. Είναι επιτακτικό κάτι τέτοιο. Ιδίω ε, στις σημερινές συνθήκες, ε, γιατί έχουμε αποθέματα τα οποία πιέζονται πάρα πολύ και χρειάζεται να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση σε επίπεδο βιοποικιλότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πατράου. Για να ολοκληρώσουμε, ο κύριος Χάντον. Thank ε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές μας. Πάντα είναι χρήσιμο να ακούμε τα πράγματα αυτά από τους ανθρώπους που έχουν άμεση εμπειρία του κλάδου και που καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη όλους αυτούς τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι προτείνουν για το μέλλον. Και βλέπω ότι υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία ανάμεσά τους, ότι όντως τα πράγματα θα πρέπει να τροποποιηθούν όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των ελευτικών πόρων στο μέλλον, παντού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αυτό είναι το εύκολο τμήμα. Συμφωνούμε για συγκεκριμένες αρχές. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι τα τρία βασικά ζητήματα των TFC των απορρίψεων και της αποκέντρωσης είναι ζητήματα τα οποία απασχόλησαν και τους τρεις ομιλητές. Και πολύ σωστά. Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι κάπως άβολα όταν Κάνουμε εδώ πέρα μια συζήτηση σαν να σχεδιάζαμε ουσιαστικά απαγόρευση των απορρίψεων βάσει των, των εκτινό, εκτιμόμενων ποσοστών απορρίψεων, όπως είπε και ο μιλητής μας στην παρουσίασή του. Στο έγγραφό του βέβαια πολύ σωστά λέει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες για να αποφύγουμε τις απορρίψεις μέσω συγκεκριμένων μέτρων. Και αυτό είναι σημαντικό σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το να επιβάλλουμε αυθαίρετα απαγορεύσεις στις απορρίψει δεν είναι ρεαλιστικό, ούτε μας βοηθάει τελικά. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να εφαρμόζονται κάποια μέτρα αποτρεπτικά ως προς τις απορρίψεις. Τώρα για τα TFCs η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τις μεταβιβόμενες αλληλευτικές παραχωρήσεις ως λύση για την ε, ικανότητα, την υπερβολική πλεονάζουσα ικανότητα αλίευσης. και λέγεται ότι αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλους τους ελευτικούς στόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να εφαρμοστεί αυτό, ιδίως διασωνηριακά θα ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και για τα αλλιευτικά αυτά έθνη τα οποία έχουν λύσει το πρόβλημα της πλεονάζωσης αλλιευτικής ικανότητας. Ποια είναι η άποψη όμως των προσκεκλημένων μας για το ζήτημα αυτό, όσον αφορά δηλαδή την υποστήριξη, τη μη υποστήριξη για τα υποχρεωτικά TFC, όσον αφορά τώρα το ζήτημα της αποκέντρωσης. Μ' άρεσε πολύ ο τρόπο με τον οποίο ο κύριο Βίσαρ σχολίασε το ζήτημα αυτό όσον αφορά την αποκέντρωση την περιφερειοποίηση και το πώ θα μπορούσε να ρυθμιστεί μέσω από την ε, συνθήκη. Όπω έχω πει και στο παρελθόν για το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν ε, τρελό να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στι ελευτικέ μα κοινότητε και να του πούμε να τι πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει στην πράξη, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε εξαιτίας της κοινοτική νομοθεσία. καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας έκανε να εμφανιζόμαστε εντελώ ε, ανόητοι. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να υποστηρίξω ένα πακέτο μεταρρύθμισης της κοινή ελευτικής πολιτικής που θα ακολουθούσε αυτό το δρόμο. Ο κύριος Βίσερ έχει απόλυτο δίκαιο όταν λέει ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις αρμοδιότητες στις απόφαση που έχουμε προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση για ένα σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη σε αντίθεση δηλαδή με πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί στα πλαίσια της κοινή ερευνητική πολιτικής μέχρι τώρα. Και αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα καταφέρουμε να κερδίσουμε και την υποστήριξη όλων των μελών των ελευτικών κοινοτήτων μας και θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε δηλαδή μία λύση ακόμα και για το ζήτημα της βιωσιμότητος, προκειμένου να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα αποθέματα και για τις μελλοντικές γενναίες. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Ο κύριος Πρόεδρος βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ανησυχεί λίγο για τον χρόνο, επομένω διατηρώ τα υπόλοιπα σχολιά μου για μια άλλη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν στι ερωτήσεις και στα σχόλια των κύριων βουλευτών. Παρακαλώ, κύριε Μαξουίν. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα ενδεχομένω ε, να ξεκινήσω απαντώντα ε, στα ερωτήματα του κυρίου Στίβενσον. Όπως είπε, νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε καλύτερα την περιφερειακή διάσταση στην ελευτική πολιτική. Κανένα πρόβλημα δεν έχω εγώ με την χρήση ενός μηχανισμού αποθήκευσης για κάποια είδη. Το κάνουμε άλλωστε αυτό. Υπάρχουν ορισμένα είδη, πελαγικά κυρίως, οι σαρδίνες, ο τόνος και άλλα, για τα οποία δεν ενδείκνυται η καταστροφή, είναι καλύτερο να αποθεκευτούν. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα οστρακοειδή. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα είδη τα οποία δεν μπορούν να καταψυχθούν, δεν καταψύχονται καλά. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αν δούμε τον τόπο των ελευτικών δραστηριοτήτων, οι περισσότεροι λιμένες, οι ελευτικοί λιμένες στην Βόρεια Ευρώπη βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποδομή κατάψυξης. Εγώ στην περιοχή της Σκοτίας που βρίσκομαι θα έλεγα ότι το πιο κοντινό μέρος απόψυξης είναι στο Αμπερντίν, που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ μακριά από το λιμένα λίευση. Για ποιο λόγο να γίνει ένα ολόκληρο ταξίδι που θα κρατήσει μία μέρα για να καταψυχθούν κάποια είδη. Επίσης, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα ασφάλισης για το ζήτημα αυτό εγώ όσον αφορά την κατοικία μου πληρώνω ένα πρόγραμμα ασφάλισης σε περίπτωση που συμβεί ένα σεισμός και πέσει το σπίτι μου. Μπορεί όμως να λειτουργήσει κάτι αντίστοιχο και στον δικό μας τον τομέα. Όταν έχουμε αλλοίς οι οποίοι δεν καταφέρουν να πουλήσουν τα αλλιεύματά τους, να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα αποζημίωσης Εργάζομαι για, από τους ε, για μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις παραγωγών στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε το έτος αλίευσης, προχωρήσαμε σε εκφορτώσεις 203.000 τόνους ε, ψαριών εκφορτώσαμε και 47 τόνοι πέρασαν, 0,01% δηλαδή περίπου πέρασαν σε αυτό το σύστημα της αποθήκευσης. Το έχουμε δει αυτό για διάφορα είδη όπως η γλώσσα. Το ποσοστό αυτό μάλλον πέρασε στο σύστημα της παρέμβασης, με συγχωρείτε, όχι της αποθήκευσης, της παρέμβασης. Πολλές φορές όμως το σύστημα αυτό δεν μπορεί να καλύψει το κόστος της παραγωγής. Η κυρία Φράγκα μας είπε ότι οι απορρίψει την πικραίνουν. Αυτό συμβαίνει και για πάρα πολλούς αλείς. Τίποτα δεν είναι πιο αποκαρδιωτικό από το να αλλιεύει κανείς, να ψαρεύει και να πρέπει να πετάει στη συνέχεια τα αλλιεύματα αυτά, ακριβώς επειδή αυτό λένε οι κοινοτικέ νομοθεσίε. Αυτό που λέμε σήμερα εδώ είναι ότι υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη στα δυτικά της Σκοτία που πετάνε γάδο, πολλά άλλα είδη ακριβώς επειδή υπάρχουν τέτοια μέτρα τεχνικά αλίευσης τα οποία μας επιβάλλουν να προχωρούμε σε απόρριψη. Δεν μας επιτρέπουν να εκφορτώνουμε αυτά τα είδη. Αν πικραίνεστε λοιπόν εσείς κυρία Φράγκα φαντάστε πόσο πικραίνονται και τι απόγνωση αισθάνονται οι ίδιοι οι αλείς οι οποίοι αναγκάζονται πραγματικά να πετάξουν πάλι μέσα στη θάλασσα τα αλλιεύματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να συντοπίσουμε ότι οι απορρίψει ουσιαστικά έχουν τρεις συνιστώσεις. Έχουμε απορρίψει εμπορεύσιμων ψαριών, για τα οποία δεν υπάρχει ποσόστοση εκφόρτωση. Σε ορισμένε περιπτώσεις όμως ε, αυτό μπορεί να πάρει και τη μορφή του high grading. Υπάρχουν ε, απορρίψει που έχουν να κάνουν... Δεν ακούγεται ο μιλητή, μας συγχωρείτε. Απορρίψεις λοιπόν πολύ νέων ψαριών που βρίσκονται κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ηλικία και μεγέθους, τα οποία δεν επιτρέπεται πάλι να εκφορτωθούν και στην περίπτωση αυτή πάλι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να δοθεί μια άδεια ακόμα και για τα νεότερα αυτά ψάρια. Καταφέραμε για το γάδο, για παράδειγμα, να περάσουμε από τα 17 μιλιμήτρες στα 120. Πολλές φορές όμως πιάνουμε και πολλά άλλα πράγματα, πολλά άλλα είδη τα οποία ζουν στο βυθό της θάλασσας. Αν πρέπει όμως να εκφορτώσουμε όλα αυτά τα είδη, τα οποία δεν είναι ψάρια, και να τα καταψύξουμε και όλες, καταλαβαίνετε ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Και ξέρετε ότι πολλές φορές όταν α, ψαρεύει κανείς με εργαλεία τέτοια αλλιευτικά τα οποία αλλιεύουν διάφορα είδη από το βυθό της θάλασσας, τότε αναγκαστικά θα πιάσει κανείς και πράγματα τα οποία δεν θέλει να αλλιεύσει. Το να χρησιμοποιήσουμε όμως από το 2013 και μετά μία ενιαία απαγόρευση τη απόρρευσης, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. οποιοδήποτε εργάζεται στον τομέα τη αλεία ξέρει ότι η απαγόρευση αυτή θα είναι στην πράξη πολύ πιο θεωρητική από ότι λειτουργική. Σαφώ θέλουμε να μειωθούν οι απορρίψει και αυτό γίνεται στην πράξη. Και αυτό που θέλω να πω, κυρία Φράγκα, είναι ότι ένα τρόπο για να μειώσουμε τι απορρίψει δεν είναι μέσω τη αγορά. Και δεν μπορεί να επιληθεί επίση κατά αυτόν τον τρόπο και το πρόβλημα της πλεονάζουσας ικανότητας αλίευσης μέσω των TFCs. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μη κατάλληλα μέτρα, κατάλληλα μέτρα προκειμένου να λύσουμε προβλήματα και στην πραγματικότητα να κάνουμε τα προβλήματα ακόμα χειρότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, παρακαλώ να είστε συγκεκριμένοι στις απάντησή σας. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ένα τρομερό παράδειγμα όπως αυτό της ε, χωματίδας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να εγκαταλείψουμε μια ολόκληρη πολιτική. Τα τελευταία χρόνια ε, ε, είδαμε τεράστια αύξηση του αποθέματος. Είναι πιο ψηλό από ό,τι ήταν τα τελευταία 50 χρόνια και τα τελευταία χρόνια ε, έχει μειωθεί η ικανότητα της, ε, ε, του, του, του τομέα κοπής των ψαριών και γι' αυτό υπάρχει αυτή η εικόνα που μας περιγράψατε. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο όλοι μάθαμε έτσι, έχει αυξηθεί η ικανότητα του το δυναμικό του τομέα κοπής των ψαριών και έτσι το πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί το 2012 και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ περισσότερη ε, χωματίδα, μπορούμε όμως να τη χειριστούμε. Απ' την άλλη είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση, διότι εάν ε, πιάζει κανείς ψάρια και τα διαθέσει στην αγορά σε πολλές χώρες ε, το, και έρθουν οι οργανώσεις παραγωγών και δεν μπορείτε να συμφωνήσετε ε, πώς θα οργανώσετε την αγορά, εάν οι Ολλανδοί δεν μπορούν να μιλήσουν με τους Γερμανούς ε, για το πώς θα πρέπει να γίνει η Ιδανή με τους Ολλανδούς, διότι οι ε, αρχές ανταγωνισμού λένε ότι αυτό γίνεται για να επηρεάσουμε τις τιμές. Αλλά δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο, το κάνουμε ε, για να ε, μπορεί να γίνει σωστή επεξεργασία των ψαριών και συμφωνούμε απόλυτα. Και όταν λέμε ότι η παρέμβαση είναι καλή, είναι καλό όταν πέντε ε, σκάφη υπάρχουν και η τιμή είναι χαμηλή και δεν είναι δίκαιο να πουλήσουν μόνο δύο από τα σκάφη τα ψάρια τους και τα άλλα τρία να μην έχουν τίποτα. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο ασφαλείας. Θέλουμε να είμαστε δίκτυο ασφαλείας, όχι για τι μεγάλε ποσότητες, και το ίδιο ισχύει ε, για την απαγόρευση, για, για, ε, για την απαγόρευση των απορρίψεων. Όλοι είναι υπέρ. Όλοι είναι υπέρ ε, της μείωσης. Δεν είναι... Ο... Όταν Όταν ένας ε, αλλιέας τη Δευτέρα ε, έχει αλλιεύσει ψάρια και πρέπει να τα απορρίψει, τα απορρίπτει, την Πέμπτη όμως ε, δεν έχει κανένα πρόβλημα παραβίαση στο κανόνα. Ποιο θέλει τώρα ο αλλιέας ή ο κανόνας και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, στην μεικτή αλλία. Δεν θα πρέπει όμως να βρούμε μια χοντρική λύση για όλα αυτά. Οι απορρίψει είναι ένα θέμα το οποίο εύκολα συζητιέται στα πάρτι, στις δεξιώσει με ένα ε, ποτήρι κρασί στο χέρι, αλλά το πρόβλημα, το πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και θα πρέπει να συνεργαστούμε για την επίλυσή του. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριος Φερνάντες, εγώ Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία στο ρόλο των οργανωσιών παραγωγών ε, και στα έσοδά του και στο θέμα των απορρίψεων. Καταρχήν, για τις οργανώσεις παραγωγών. Και όπως είπε και η κυρία Φράγκα, έχουμε οργανώσεις ε, μεγαλύτερε και οργανώσεις ε, πιο μικρές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, στην Πορτογαλία ένα σκάφος στα τρία συμμετέχει σε οργάνωση παραγωγών. Αλλά Α, δηλαδή μιλάμε για το 33%. Αλλά αν ε, μιλούσαμε για τον τομέα της Σαρδέλας, 92-93% των σκαφών συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών. Ποιος έχει τώρα λοιπόν καλύτερα έσοδα, όσοι είναι εντός ή εκτός των οργανώσεων παραγωγών τουλάχιστον ε, για τη χώρα μου, αυτοί που συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών. Έτσι λοιπόν, η πρώτη πρόκληση που τίθεται είναι να δημιουργηθούν οι προποθέσει για να ενισχύσουμε τις οργανώσεις παραγωγών και να έχουν μεγαλύτερα δικαιώματα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί παρέμβασης. Μπορεί να είναι ε, πιο απλουστευμένοι, ε, ούτε σε μένα βέβαια φαίνεται σωστό να φτάνουμε ε, σε καταστάσεις ε, όπου πετάμε εκτός ε, τα ψάρια. Δηλαδή να τα ξαναρίχνουμε στα λασσά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να το υποστηρίξουμε, αλλά Πρέπει επίσης εδώ να μην ξεχνάμε μια ουσιαστική πτυχή. Ο ξεχρονισμός και η διαγωνιστικότητα και η καινοτομία του τομέα απαιτεί οργανώσεις, παραγωγούς και μηχανισμού παρέμβαση. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς θα γίνει η ανανέωση ενός σκάφους, εξυγχρονισμός ενό σκάφου και να, για να πληρούνται καλύτερα ε, οι προποθέσει ασφαλεία και να ε, μπορεί να υπάρχει καλύτερη ποιότητα στη μεταποίηση. Ε, αν δεν υπάρχουν περισσότερα έσοδα, επίσης ε, ε, και για το πλήρωμα ε, πρέπει να περάσουμε μέσα από του οργανώσει παραγωγών. Η κυρία Πατρέων αναφέρθηκε εδώ ε, στι διεπαγγελματικέ οργανώσει. Επιτρέψτε μου και στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια. Τα τελευταία 10-15 χρόνια είδαμε μία αλλαγή του τρόπου που φτάνουν τα λευτικά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή. Σήμερα οι δομές ε, της διανομής, ε, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν ε, καταψυγμένα προϊόντα, αλλά έχουν και νοπά προϊόντα και επίσης έχουν και προϊόντα το καλλιέργεια, σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενα, αλλά έχουν και τέτοια προϊόντα και νοπά και καταψυγμένα πριν 10-15 χρόνια στην Πορτογαλία τουλάχιστον. Αυτό δεν υπήρχε σποραδικά. Βλέπω μία μέρα την εβδομάδα είχαμε αλευτικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν ε, αυτή η δομή ε, διανομής υπερισχύει σήμερα και πρέπει ε, και επίσης καθώς ε, προσφέρουν στον καταναλωτή προϊόντα όλα τα χρόνια πρέπει να μπούμε σε μία διαπραγμάτευση Τρίτο σχόλιο, σε ό,τι αφορά τι απορρίψει, Θα ξαναναφέρω την προειδοποίηση που έκανα στην αρχή, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, όπως σα είπα. Η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι υπερβολικά βολιταριστική, γιατί το θέμα είναι το εξή Οι απορρίψει είναι θέμα χρονοδιαγράμματος, είναι θέμα timing. Οι απορρίψει ε, θα ε, σημαίνουν ότι θα ε, πρέπει να υπάρχει περισσότερη δουλειά επί του σκάφους. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται διαλογή των ψαριών ε, για το ποια θα εκφορτωθούν και ποια θα απορριφθούν. Και σε όλη και σε όλη την αλυσίδα. Δηλαδή δεν αρκεί να πούμε α, αυτά είναι για εχθιάλευρα, γιατί όσο είναι για εχθιάλευρα ε, πρέπει να μεταπηθούν με διαφορετικές ε, προϋποθέσεις από τα ψάρια που, προδε... που οδεύουν για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν μπορούμε να τα μπλέξουμε αυτά. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μία σειρά προϋποθέσεων σε έναν ολόκληρο τομέα για να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Εκτός αν θέλουμε να έχουμε ένα είδος ε, fast code. Και επίση ε, είδαμε τι έκανε και η Νορβηγία, αλλά η Νορβηγία χρειάστηκε 20 χρόνια. 20. Και κατόπιν η Νορβηγία έχει μία δομή ε, πολύ αναπτυγμένη σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή χρησιμοποιεί πολύ τέχθη άλευρα για την υδατοκαλλιέργεια αν ε, δεν χρησιμοποιηθούν ε, αυτά τα ψάρια, αν πάνε για καταστροφή, θα προσπαθήσουν οι αλληλείς να δημιουργήσουν μια παράλληλη αγορά, γιατί η καταστροφή δεν τους δίνει εισόδημα. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε εδώ μια επικοδομητική προσέγγιση, δεν μπορούμε να έχουμε επιβολή. Γιατί αν ε, μιλάμε μόνο για επιβολή, όπως σας είπα, είναι πολύ βολονταριστική η θέση της Κομισιόν και δεν έχουν ληφθεί υπόψη ή αλήθεια. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να έχουμε μια πιο στιαδιακή εισαγωγή αυτού του μέτρου και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θέματα που έχουν θέσει και μεγάλες οργανώσεις ε, παραγωγών, όχι μόνο οι μικρές οργανώσεις που υπάρχουν στη χώρα μου λόγου χάρη, έχουν θέσει θέματα πρακτικά οι οργανώσεις αυτές, δηλαδή πώς στην πράξη θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα των απορρίψεων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο πάνελ και να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέμβασή σας, για τις παρεμβάσεις σας και να αλλάξουμε τώρα εδώ θέση, να έρθουν οι προσκεκλημένοι του δεύτερου πάνελ και θα αρχίσουμε σε 2-3 λεπτά. την κυρία Señorías, Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο πάνελ, αφού ξεκουραστήκαμε και λίγο. Θα αλλάξουμε, όπως σας είπα, τη σειρά των ομιλητών και θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της κυρίας Γκέρλινγκ. Έχετε το λόγο. Για δέκα λεπτά, όπως είπαμε και πριν.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 Adelante. Good afternoon, ladies and... Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ζήτω συγγνώμη που δεν ξεκινήσαμε αμέσω, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Λέγομαι Τατιάνα Γκέρλινγκ. Εκπροσωπώ το ε, Διεθνέ Ταμείο για τη Φύση, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση και εκπροσωπώ ε, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αλληλείας, ε, τη λεγόμενη Πρωτοβουλία Εφιούς Αλληλείας, Smart Fishing Initiative. Προσπαθούμε να πετύχουμε αποτελέσματα μόχλευσης για να βελτιώσουμε τη διαχείριση της αλληλείας σε όλο τον κόσμο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το εμπόριο του κορέγονου ε, την διαχείρισή του και ιδιαίτερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας στην διαχείριση και το εμπόριο του κορέγονου. Όπως ε, μίλησαν οι προλαλήσαντες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την εισαγωγή ε, ηχθείων και θαλασσινών. Το 60% των ψαριών που καταλήγουν στο πιάτο καταναλωτή δεν προέρχονται από ευρωπαϊκά ύδατα, προέρχονται από άλλες χώρες. Και η Κίνα παίζει σημαντικό ρόλο θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ε, δείξω από πού έρχονται τα ψάρια και τι γίνεται με αυτά. Λίγα λόγια για τον κορέγονο. Το μεγαλύτερο μέρος ε, του κορέγονου προέρχεται όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τον Βόρειο Ειρηνικό και την και τον βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό. 7, πάν, 7 εκατομμύρια τόνοι παράγονται σε όλο τον κόσμο, περίπου το μισό ε, αποτελείται από γάδο και ε, μπακαλιάρο της Αλάσκας. Ε, οι συνολικέ εκφορτώσεις τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής το 2009, σύμφωνα με τι στατιστικέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι. Για να έχετε μια ιδέα του μεγεθού του τομέα. Τι γίνεται λοιπόν με τα ψάρια αυτά τα περισσότερα, ιδιαίτερα τα ψάρια από την ε, Ρωσία, καθώς και η ρωσική αλληλεία μπακαλιάρου της Αλάσκας ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο, περίπου το ίδιο ο ίδιος όγκος ε, αλλιεύεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, στις, στις ακτές της Αλάσκας και περίπου 1.900.000 τόνοι προέρχονται από την θάλασσα Μπάρεντ. Ο μεγαλύτερος όγκος των ψαριών πηγαίνει στην Κίνα για μεταποίηση. Η πρώτη εικόνα που είδατε είναι μια εικόνα, ε, μια φωτογραφία που πήρα σε ε, Κινέζικο Εργαστήριο μεταποίηση πριν δύο μήνες. Ε, η Κίνα δεν έχει δικό τη στόλο για αλληλεία κορέγονου. Εξάγει όμω τα προϊόντα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Αμερική και όλο και περισσότερο στη Βραζιλία. Ο μιλητής του πρώτου, ένας του πρώτου πάνελ ανέφερε την μείωση των τιμών για τον Κορέγονο και την ε, εισαγωγή τέτοιων νυχθείων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη συνεργασία με τους ε, Κινέζους ε, μεταποιητές θα ήθελα να σας πω ότι η Βραζιλία έχει όλο και περισσότερο όρεξη για τέτοια προϊόντα και η ίδια τάση διαπιστώνεται και στην εσωτερική, συνεχόρια κινέζικη αγορά. Να σας δώσω μια εικόνα, έναν υπολογισμό ε, σχετικά με τον ε, δρόμο ε, που ακολουθεί ο Πακαλιάρος της Αλάσκας για να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά από τη Ρωσία Μικρό ποσοστό φτάνει κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο μέρο των ψαριών φτάνει στην Ευρώπη μετά μέσω των Κινέζων μεταποιητών. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε την ε, αλυσίδα από το σκάφος ε, στους μεταποιητές, στους ε, μεταφορείς που καταλήγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο, το πιστοποιητικό προέλευσης που εισήχθη από, την, από τον κανονισμό IUU για την αλληλεία απλά στις αρχές του 2010. Απαιτείται λοιπόν πιστοποιητικό για κάθε ε, εξαγωγή ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ως περιβαλλοντική οργάνωση εξετάσαμε το ρόλο που παίζει το πιστοποιητικό ε, στο να διασφαλίζει να μην καταλήγουν στην ευρωπαϊκή αγορά παράνομα ψάρια. Μετά από την επισκόπηση αυτή διαπιστώσαμε δύο σειρές θεμάτων που συνδέονται με το πιστοποιητικό. Καταρχήν ο κανονισμός ε, IUU, για την αλία απλά δηλαδή, παράνομη λατρεία και άναρχη αλία, ε, ήταν το πρώτο ε, μέρος ήταν ένας ε, κανονισμός που αφορούσε κάθε ε, αλλιέα. Δεν ε, είναι κανονισμός ο οποίος αφορά μόνο κάποια υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης. Είναι κάτι που αφορά κάθε επιχείρηση. Αλλά πρέπει, είναι αυτό το σύστημα επαρκές, υπάρχουν σαφείς κανόνες και κριτήρια. Η επαλήθευση είναι, γίνεται πράγματι σωστά και ε, ξέρω ότι ο επόμενος ομιλητής ε, θα αναφερθεί στο θέμα αυτό. Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι οι εξαγωγείς είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν με αυτόν τον κανονισμό. Έχει γίνει αρκετή δουλειά ώστε να εξηγηθεί στις ε, χώρες εξαγωγής πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Άλλη ερώτηση είναι εάν υπάρχει απαραίτητη υποδομή ώστε τα πιστοποιητικά αλληλείας πράγματι να λειτουργούν και να παίζουν το ρόλο που πρέπει. Υπάρχουν ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το εμπόριο του κορέγονου και την ε, ε, διασφάλιση της ε, βιώσιμης αλληλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την εισαγωγή καινοτόμου ε, συστήματος πιστοποιητικών αλληλείας. Μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες, ωστόσο οι άλλε χώρε ε, κοιτάνε ακόμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουν την απόδειξη ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, και να εφαρμοστεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει άλλου κανόνε και κανονισμού που μπορεί να διασφαλίσει την ε, λειτουργία του κανονισμού IUU. Ε, και δεν μιλάμε για πιο πολλά πιστοποιητικά ή πιο πολλές ανακοινώσεις, αλλά με βάση τις εμπειρίες των εξαγωγέων ε, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μαθήματα, αυτά που έμαθαν οι άνθρωποι του τομέα για να δημιουργήσει ε, κατάλληλα εργαλεία ώστε να ε, φροντίσει να μην εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά ε, παράνομα προϊόντα. Και θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ε, Κίνας. Βλέπουμε εδώ πέρα παράδειγμα από τη Ρωσία. Είτε κατευθείαν από τα ρωσικά τα φτάνει το ψάρι στην Κίνα για μεταποίηση, είτε μέσω εμπόρων που συνήθως είναι Κορεάτες. Ε, γενικά ο έλεγχος στην Κίνα γίνεται από μία αρχή στο Πεκίνο. Μπορεί ε, να φαίνεται δύσκολο δεδομένου του μεγέθους του τομέα ε, θαλασσινών στην Κίνα ε, μπορεί να φαίνεται πολύ πλοκό το σύστημα αυτό με τη μία αρχή, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του συστήματος στην Κίνα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να βελτιώσει τη ρύθμιση, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνο μία χώρα και μία αρχή που ασχολείται με ε, τα ε, πιστοποιητικά αλλιέ από πολλές χώρες. η, Ευρωπαϊκή, η, η Κίνα αποτελεί παράδειγμα για πολλέ χώρε του κόσμου, ιδιαίτερα για την Ασία και με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς θαλασσινών. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλω να σας στείλω σήμερα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές θαλασσινών το να ασχολούμαστε μόνο με την αλληλεία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει απάντηση ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη αγορά και ε, να διασφαλίσουμε επίση την προμήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψάρια για τι επόμενε δεκαετίες. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την εισαγωγή νέων συστημάτων όπω είναι το σύστημα των πιστοποιητικών αλληλεία. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν βελτιώσει, ώστε να ε, διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματο. και να μπορέσει να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες. Και τέλος, η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας είναι ο τρόπος να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά αυτόν τον κανονισμό και να διασφαλίσουμε ε, τα, ε, ε, την αγορά ψαριών στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Και δεν θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να γίνουν διμερώς αποκλειστικά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κίνα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετάσχει και ο τομέας θαλασσινών και άλλοι δημόσιοι φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία του κανονισμού που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάρτισον τώρα έχει το λόγο και 10 λεπτά παρακαλώ. Yes, good evening to every one of you. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ, με, σας ευχαριστώ πολύ για την καταπληκτική ευκαιρία που μου δίνετε να αποταθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Θα μιλήσω σήμερα για τις μοριακές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ψευδούς σήμανσης. Νομίζω ότι α, υπάρχει το ζήτημα αυτό πάρα πολύ καλά στο γενικότερο ζήτημα το οποίο συζητάμε, δηλαδή τα ποιοτικά προϊόντα λίας και τα οποία πηγαίνουν προς τους καταναλωτές. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω πώς οι μοριακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την ιχνηλασιμότητα των αλλιευμάτων και των προϊόντων αλίας. Πρέπει να πάμε πιο μακριά, πέρα από τη σήμανση και την απλή πιστοποίηση. Τα δύο αυτά ζητήματα τα αναφέραμε σήμερα και πιστεύω ότι οι μοριακέ τεχνολογίε μπορούν να μα επιτρέψουν να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Σαφώ υπάρχουν κάποιε ευκαιρίε που προκύπτουν από τι μοριακέ τεχνολογίε. Πολύ συχνά υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μιλάνε για τι νέε τεχνολογίε και τι δυνατότητε που μα δίνουν για την καλύτερη επιτήρηση και παρακολούθηση της αλίας οι μοριακές όμως τεχνολογίες και οι γενετικοί δεν αναφέρονται αρκετά συχνά. Αυτό είναι κρίμα. Δεν θα μιλήσω για την παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία, άλλωστε η Επιτροπή σας πρόσφατα δημοσίευσε μια σχετική έκθεση. Πέρα όμως από την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλλία, υπάρχει και το πρόβλημα της ψευδούς σήμανσης. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να εντοπίσουμε το φαινόμενο αυτό και σαφώς θα πρέπει να προστατεύσουμε τον καταναλωτή από αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν πάρα πολλά δελτία τύπου τα οποία τα βλέπετε, δημοσιεύτηκαν σε διάφορες εφημερίδες και όπως βλέπετε κάτω αριστερά πολλές φορές η ψευδής σήμανση μπορεί να έχει πολύ επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι συστήματα ηχνερασιμότητας που έχουμε μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όσον αφορά την πληροφορία, την ενημέρωση προς τον καταναλωτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο καταναλωτή μπορεί να δραματίσει και αυτός ένα σημαντικό ρόλο προκειμένου να καταφέρει να διαμορφώσει προς όφελός του την διαχείριση της αλίας. Να αναφερθώ για παράδειγμα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μια σχετική ιστοσελίδα που μπορεί πραγματικά να σας ενημερώσει για το τι μπορούμε να κάνουμε με την αλληλεία πέρα από κάποιες απλές συνταγές που βλέπουμε. Όσον αφορά το ζήτημα της εχνελασιμότητας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ήδη μια κοινοτική νομοθεσία. Για παράδειγμα έχουμε τον κανονισμό 178-2002, ο οποίος θέτει πολύ αυστηρούς κανόνες σήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα αλίας. Επίσης έχουμε και τον νέο κανονισμό για την επιτήρηση της αλλιευτικής πολιτικής αναφέρεται και αυτός ο καονισμός στην εκλασιμότητα και έχουμε βέβαια και τον καονισμό για την παράνομη και λαθρέα αλία που και αυτός με τη σειρά του έχει συμβάλει στο να εξασφαλίσουμε ότι τα ψάρια τα οποία αγοράζουμε έχουν ε, αλλιευθεί νόμιμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν, ε, παράνο, έχουν ε, ανάλογη νομοθεσία όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση των προϊόντων αλίας. Πολύ καλά λοιπόν όλα αυτά, αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε ένα σύστημα εχνηλασιμότητας το οποίο να μας επιτρέπει να ελέγχουμε κάθε στάδιο της, από την αλίευση μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος αλίας. Όπως σας είπα, μέχρι στιγμή στηριζόμασταν μόνο σε δύο μέσα, σήμανση και πιστοποίηση. Χρειαζόμαστε όμως και κάποια ανεξάρτητα μέτρα ελέγχου και νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν οι μοριακές τεχνολογίες ιδανικά αυτά τα ανεξάρτητα μέσα ελέγχου θα έπρεπε να απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις. Για ποια είδη μιλάμε, από πού προέρχονται τα προϊόντα αλίας και θα μπορούν επίσης να μας βοηθούν να διακρίνουμε ανάμεσα σε προϊόντα λίας και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Ευτυχώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γενετική, το DNA, προκειμένου να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους χημικούς δείκτες οι οποίοι μας επιτρέπουν να δούμε ποια είναι η ακριβής προέλευση κάποιων προϊόντων. Όλοι μας φέρουμε μέσα μας ένα DNA, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τον κώδικα της ζωής και είναι αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί τον έναν από τον άλλον. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά, για παράδειγμα, από την αστυνομία τα δεδομένα DNA. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως τη γενετική, των DNA, προκειμένου να καταφέρουμε να διαφοροποιήσουμε, για παράδειγμα, ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές περιοχές της γης και κατ' επέκταση ψάρια τα οποία προέρχονται από διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές. Και θα μπορούσε το DNA να χρησιμοποιηθεί και σαν δείκτης, προκειμένου να διαφοροποιηθούν κάποια είδη στον τομέα της μεταποίησης. Υπάρχουν πλέον γενετικοί δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ταυτοποιήσουμε κάποια μεταποιημένα προϊόντα, για να δούμε δηλαδή για ποια ψάρια ακριβώς μιλάμε, για ποια είδη ακριβώς μιλάμε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή συγκεκριμένε γωνιεδιακές αλληλουχίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τον κλάδο της αλίας προκειμένου να έχουμε καλύτερα συστήματα εχνηλασιμότητας. Μια μεγαλύτερη πρόκληση είναι το να καταφέρουμε να απαντήσουμε στο έρχεται το λευτικό προϊόν το οποίο καταναλώνω. Για πάρα πολύ καιρό πιστεύαμε λόγω του ανοιχτού χαρακτήρα της αλίας ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τα είδη και θεωρούσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και γενετικούς δείκτες γι' αυτό. Πρόσφατα, σε μια έρευνα που έγινε, είδαμε ότι ε, υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι γενετικοί πληθυσμοί όσον αφορά συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένε περιοχές, για παράδειγμα ο γάδο του Ατλαντικού. Και είδαμε ότι υπάρχουν όντως γενετικές διαφορές ανάμεσα στον γάδο της Βαλτική ή τον γάδο της Μεσογείου. Αυτό φαίνεται συγκεκριμένα στην εικόνα που βλέπετε, στην πάνω εικόνα στη διαφάνεια, όπου βλέπετε ότι με διαφορετικό χρώμα έχουμε διαφορετικά είδη. Όσο πιο συγγενή είναι τα χρώματα στην εικόνα, τόσο πιο κοντά από γονιδιακής πλευράς είναι τα είδη τα οποία βλέπετε να απεικονίζονται. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λοιπόν το δεδομένο αυτό από τι αρμόδιε αρχέ προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώ από πού προέρχονται κάποια είδη. Για παράδειγμα βλέπετε κάποια είδη τα οποία παρουσιάζουν γενετικά χαρακτηριστικά τη Βαλτική θάλασσα. Μπορούμε να, Μπορούμε να πάρουμε ιστό από τα ψάρια αυτά, να γίνει μια γονιδιακή ανάλυση και να εντοπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον χώρο, τη θάλασσα προέλευση των ψαριών αυτών. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πολύ μεγάλο δειγματολόγιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νοπά, κατεψυγμένα ψάρια, μαγειρεμένα ψάρια, ψάρια τα οποία περιέχονται σε κάποια κονσέρβα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δείχτες αυτούς ακόμα και σε τηγανισμένα ψάρια ή ακόμα και σε κονσέρβες που περιέχουν πολλά διαφορετικά είδη. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες αυτές, όπως σας είπα, για την παρακολούθηση, για την επιτήρηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί γίνονται όλο και πιο δημοφιλή διάφορα συστήματα πιστοποίησης. Το DNA όμως και η γενετική γενικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταφέρουμε να δούμε ποιον δρόμο έχει ακολουθήσει ένα προϊόν, από την αλίευση μέχρι την κατανάλωση. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε την γενετική και στα πλαίσια ενός γενικότερου πλαισίου επιστημονικής ανάλυσης, αν πρέπει για παράδειγμα κανείς να κάνει μια προσφυγή στο δικαστήριο και να πρέπει να καταθέσει κάποια πιστήρια, κάποια επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πιστήρια. Είναι πολύ σημαντικό όμω να καταφέρουμε να έχουμε και τα απαραίτητα μέσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα επιστημονικά αυτά δεδομένα κοστίζουν πολύ πιο ακριβά από την απλή ανάλυση που μπορεί να γίνει βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη επανάσταση όσον αφορά την γενετική. Μας δίνονται πολύ περισσότερες ευκαιρίες και πιστεύω ότι θα πρέπει να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες αυτές. Βλέπουμε ότι οι γονιδιακές αναλύσεις, οι αναλύσεις αλληλουχίας του DNA παρουσιάζουν όλο και χαμηλότερες τιμές. Η τάση αυτή είναι συνεχής. Επίσης, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η αλληλουχία του DNA ως αποδεκτικό στοιχείο. Έχουμε επίσης διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως η βάση δεδομένων Fishball. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια γενικότερη δομή γενετικού πληθυσμού θαλασσίων ψαριών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όλο και περισσότερο. Και έχουμε βέβαια και διάφορα λογισμικά, αναλυτικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο από τους επιστήμονε και είμαστε πλέον σε θέση να συνδυάσουμε παρα... γενετικές παραμέτρους με περιβαλλοντικές παραμέτρους, προκειμένου να κάνουμε μια καλύτερη ανάλυση. Πολύ καλό όλα αυτά, αλλά πόσο κοστίζουν και πραγματικά αξίζει να κάνουμε αυτή την επένδυση. Για να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Η ανάλυση αυτή έγινε από διάφορα Ινστιτούτα τα οποία θα μπορούσαν παγκοσμίως να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά τη νέα αυτή γενετική ανάλυση. Του ζητήσαμε λοιπόν να κάνουν γενετική ανάλυση όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων αυτών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε όλες αυτές τις έρευνες που γίνανε σίγουρα το όφελος ήταν πολύ σημαντικότερο από το κόστος. Πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί η μελέτη αυτή και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από όλου του εμπλεκομένου στον κλάδο τη αλεία. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε πραγματικά να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Στι διαφάνειε βλέπετε πάρα πολλά παραδείγματα όπου έχει χρησιμοποιηθεί η γενετική σε διάφορα προγράμματα εχνηλασιμότητα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα όπου έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία τα δεδομένα μάλλον DNA, προκειμένου να επιβληθεί ο νόμος, είτε για την ποστοποίηση, είτε για την ταυτοποίηση της προέλευσης, τόσο για ελεύθερα είδη ή για είδη εκτροφής. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι όλο και πιο διαθέσιμες τεχνολογίες αυτές, αυτέ. Θα πρέπει τα γενετικά δεδομένα να συλλέγονται, να είναι διαθέσιμα σε μια βάση δεδομένων προς όλους τους τελικούς χρήστες. Πρέπει να καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε τα εργαστήρια αυτά, τα οποία υφίστανται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν όμως πολλές αρμόδιες εθνικές αρχές που γνωρίζουν την ύπαρξη των εργαστηρίων αυτών. Χρειαζόμαστε επίση την απαραίτητη επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορε νομικέ προσφυγέ που γίνονται. Όσον αφορά τώρα την συλλογή των δεδομένων από του ερευνητέ, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και του ερευνητέ αυτού, του επιθεωρητέ, με συγχωρείτε, προκειμένου να είναι σε θέση να συλλέγουν και να αναλύουν τα δεδομένα αυτά με τον κατάλληλο τρόπο. Βλέπουμε επίσης ότι οι ικανότητες αυτές για τη γενετική ανάλυση θα αυξηθούν στα διάφορα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να μπορούμε να βασιζόμαστε όλο και περισσότερο σε αυτές τις τεχνολογίες. Από επιστημονικής λοιπόν πλευράς η ταυτοποίηση των ειδών μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση του DNA και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται όλο και πιο συχνά. Η γεωγραφική προέλευση τώρα βάσει γενετικών δικτών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί Πρέπει όμως να γνωρίζουμε στην περίπτωση αυτή ποιες νομικές, ποια νομικά ζητήματα θέλουμε να διευθυντήσουμε. Αν όμως οι πολιτικοί, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, θεωρούν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την, το δρόμο αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους επιστήμονες να κάνουν μια μεγαλύτερη έρευνα σε αυτό το τομέα. Όπως σας είπα υπάρχουν πολλά εργαστήρια ήδη σε διάφορες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό και θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα εργαστήρια και θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Οι δαπάνε όσον αφορά την ανάλυση DNA μειώνονται όλο και περισσότερο και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την μειωτική αυτή τάση των τιμών. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι για να κάνουμε μια γενετική ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει να έχουμε και τι απαραίτητε υποδομέ σε τοπικό επίπεδο. Αυτά είχα να σας πω. Είμαι στη διάθεσή σας. Βλέπετε και τα στοιχεία μου. Ε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου προκειμένου να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μάρτινσον και τέλος θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Bueno, muchas Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω να μου συγχωρήσετε την, άγνα, την άγνοιά μου, γιατί <laughs> βλέπω οι υπόλοιποι συνάδελφοι ε, έχουν τόσες πολλές γλώσσες. Ε, εγώ εργάζομαι και σε τεχνικό επίπεδο στην ε, άκρη στη γωνιά της Ευρώπης, την πιο νότια γωνιά της Ευρώπης, στα στενά του Γιβραλτάρ. Και σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα και μπορώ να μοιραστώ την ε, μικρή μου εμπειρία μαζί σας. Εγώ εκπροσωπώ το μικρό στόλο που δραστηριοποιείται σε αυτή τη ζώνη από το Κονίλιο Δελαφροντέρα μέχρι το Γιβραλτάρ και στην περιοχή μου ε, δεν είναι ικανοποιημένη η Αλής ε, τελευταία με την ε, απόφαση που ληφθεί από το Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου αλλά παρόλα αυτά κατανοούμε ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να τους ικανοποιούν πάντοτε όλους αλλά θα θέλαμε κάποια μέρα, όχι μακρινή, μία επιτροπή αυτού του Κοινοβουλίου που να αποτελείται από εκπροσώπους του πιο βόρειου τμήματος που μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο πολύ τα του Νότου να έρθουν και να γνωρίσουν και τη δική μας εμπειρία στον τομέα της Αλίας, στην Κάντιθ. Ε, έχουμε αυτό τον τονισμό όταν ε, μιλάμε. Έτσι λοιπόν ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν είμαι δυσνόητος. Έχουμε δύο παραδείγματα. Εγώ προέρχομαι από το Κονίλ, από την οργάνωση παραγωγών και δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αυτή η οργάνωση παραγωγών έχει τη βάση της ε, σε μία ένωση αλλιέων ε, που είναι ένα είδος οργάνωσης διαφορετική από αυτού που γνωρίζετε. Είναι χαρακτηριστική της Ισπανίας η οργάνωση αυτή. Και Βέβαια, να σας πω ότι όχι μόνο η Ισπανία χρειάζεται να εξευρωπαϊζεται, αλλά πολλές φορές ε, χρειάζεται να ισπανοποιείται και η Ευρώπη. Και έχουμε και κάποια κέντρα ε, ελέγχου της Αλίας που ονομάζονται ηχθιόσκαλες αγορές των ηχθείων. Έτσι λοιπόν ε, θα μιλήσω για το στόλο στο Κονίλ. Βλέπετε ότι μιλάμε για ένα παραδοσιακό, για ένα στόλο, τα σκάφη. Είναι το πολύ 15 μέτρα και ε, χρησιμοποιούν ε, το αγκίστρι και χρησιμοποιούν και τα πλάδια δίχτυα, ανάλογα με τις ε, εποχές του χρόνου. Επίσης, βλέπουμε σε αυτό το διάφθαρη διαφάνεια ότι η ετικέτα από τη βάρκα μέχρι το τραπέζι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον παραδοσιακό στόλο. Γιατί οι ελείς ε, προσέχουν πάρα πολύ ε, το προϊόν καθώς πρόκειται για παραδοσιακή δραστηριότητα. Και εδώ μπορούμε να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των στόλων που φαίνεται ότι σήμερα παίρνουν ε, αυτή την ονομασία ε, παραδοσιακή στόλη δηλαδή, αλλά είναι πολύ πιο μεγάλη. Ενώ ο δικός μας στόλος είναι πράγματι πολύ μικρός. Μόνο ε, οι παραδοσιακοί αλληλείς μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα επειδή προβαίνουν στη μεταποίηση των ψαριών επί του σκάφους. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε η κοινή οργάνωση αγοράς να λάβει υπόψη ε, ότι όσο περισσότερες πληροφορίες δίνουμε στον καταναλωτή τόσο το καλύτερο και η ημερομηνία της αλίευσης ε, είναι κάτι θεμελιώδες για αυτό το μικρό στόλο. Σε αυτή την τρίτη διαφάνεια θέλω να μιλήσω για την εμπειρία του Κονίλ που πιστεύω ότι αποτελεί μια εγγύηση για τον καταναλωτή. 11 είδη που αλλιεύονται με παραγάδι. Ε, σε αυτά τα 11 είδη βάζουμε ε, την ετικέτα ο κάθε ελέας το βάζει την ετικέτα με τα ίδια του τα χέρια. Έτσι λοιπόν διασφαλίζουμε την ανιχνευσιμότητα από τη στιγμή της αλλιεύσης μέχρι να φτάσει το προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Η είναι αυτοί ακριβώς που βάζουν αυτές τις ετικέτες ε, στα ψάρια υπό αυστηρό έλεγχο για να εγγυηθούν ε, την έξτρα ποιότητα του προϊόντος ε, που πολλούνται σε αυτές τις εχθιόσκαλες. Στην ταρίφα μπαίνει η ετικέτα μόνο σε ένα είδος στο πελαγίσιο λιθρίνι. Έχουμε ένα μοναδικό σχέδιο διαχείρισης που εγώ νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα και είχε και τα περισσότερα ωφέλη. Δυστυχώς, ε, καθώς πρόκειται για μια, πρόκειται για μια πολύ μικρή ζώνη τα στενά του και υπάρχει ανταγωνισμός ε, των στόλων και από τις δύο όχθες. Δηλαδή έχουμε και ανταγωνισμό και από τους μερακινούς. Ε, και αυτοί οι δύο στόλοι εργάζονται και οι ε, και δύο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή περιοχή και ε, από την Ταρίφα βλέπει απέναντι την Ταγέρη και από την Ταγέρη φαίνονται τα παράθυρα και οι στέγες στην Ταρίφα. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πολύ στενό χώρο πρέπει να συμβιώσουν και οι δύο στόλοι και όταν οι Ευρωπαίοι έχουμε έναν αυστηρό έλεγχο και ένα σχέδιο διαχείρισης ε, της αλίας ε, για το πελαγίσιο λιθρίνη, από την άλλη πλευρά οι Μαροκινοί δεν το έχουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συναντάμε. Εκτός ε, και αν ε, είμαστε κάπως πιο έξυπνοι και αρχίζουμε να εργαζόμαστε για το καλλιέργεια, τότε αυτό το είδος θα εξαφανιστεί πολύ σύντομα. Και πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες για να μην συμβεί κάτι τέτοιο και εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτό το κατακλυσμό και αυτό όχι γιατί δεν έχουν γίνει προσπάθειες από τη δική μας πλευρά της όχθης, από τη δική μας όχθη. Η ετικετοθεσία απαιτεί καταρχήν Μάλλον διορθώνει ο μιλητή. Ε, η τα αποτελεί μια εγγύηση και έχουμε μια διαδικασία εχνηλασιμότητα που παρέχει πάρα πολλέ πληροφορίε. Το σημαντικό είναι να φτάνουν οι πληροφορίε αυτέ ε, μέχρι το τραπέζι. Η Και για να γίνει κάτι τέτοιο. Χάθηκα, λέει ο μιλητή. Μου διέφυγε μια διαφάνεια. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι γίνεται με τις παρτίδες. Με τις παρτίδες των ψαριών ε, όπου δεν ε, βάζουμε μονομένες ετικέτες και ανησυχούμε τι κάνουμε με αυτές τις παρτίδες ψαριών, τι μπορούμε να κάνουμε. Για να μπορέσουμε να διαιρέσουμε σε μικρές ομάδες ε, αυτά τα ψάρια. Όταν ε, κάποιος πάει στην καλά στον πιστηριασμό μπορεί να αγοράσει το σχάρι ένα κιλό ηχθείων και μαζί θα πάρει και όλο το έγγραφο, το αναλυτικό έγγραφο της εχνησιμότητας. Είναι, ε, μάλλον, ξεχνάμε ότι η τιμή ε, στα ψάρια δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια η τιμή της πώληση, ενώ το κόστος της συσκευασία και της ετικετοθεσίας έχει ανέβει σημαντικά. Υπάρχει λοιπόν συνεχή ζημία για τον, ε, για τον, για τον αλία, με συγχωρείτε. Έτσι λοιπόν η βιωσιμότητα είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και την κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα, γιατί αν μείνουμε χωρίς αλίες, τι θα κάνουμε. Και δεν ε, μπορούμε να εξάγουμε τα πάντα, πρέπει να διαφυλάσσουμε και την ποιότητα και πρέπει να είμαστε και λογικοί. Αλλά ούτε μπορούμε τελικά ε, και να σπαταλούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να είμαστε και κάπως πιο έξυπνοι σε όλα αυτά. Αυτές οι μικρές ε, παρτίδες είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι, σε αυτό πρέπει να δώσουμε απάντηση. Πρέπει να εργαστούμε όλοι πάρα πολύ σοβαρά προς αυτή την κατεύθυνση για να μην διαταραχθεί η εμπορική αλυσίδα. Και όπως σας είπα, τα στοιχεία από την ηχθειόσκαλα βγαίνουν με ακρίβεια όμως το πρόβλημα έγκυται ε, στη συνέχεια, στη συσκευασία. Ε, δηλαδή όλη η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι να φτάσει το προϊόν από την ηχθειόσκαλα στο τελικό καταναλωτή. Ίσως και η μοριακή επιστήμη να μας βοηθήσει. Να μπορέσουμε να βάλουμε ίσως ε, κάποια μικροτσίπ ε, στα ψάρια. Να μας επιτρέψει αυτό, να βρούμε τη λύση. Εγώ δεν ξέρω τελικά τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι δύσκολο. Θέτουμε πάρα πολλά θέματα εδώ και εγώ σας εγγυώμαι ότι ως οργάνωση παραγωγών ε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση. Αλλά πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα μικρά ψάρια. Και είναι πολλά. Και να ολοκληρώσω λέγοντα ότι ακριβώ η ετικετοθεσία είναι η ετικέτα, είναι η μεγάλη εγγύηση που προσφέρεται στον καταναλωτή και οι πληροφορίες που δίνονται στον καταναλωτή όσε και να είναι, πάντοτε δεν φτάνουν. Όσο περισσότερα ξέρει ο καταναλωτή, τόσο καλύτερο. Γιατί ο καταναλωτή έχει το δικαίωμα να μπορεί να γνωρίζει τι τρώει. Πού ξοδεύει τα χρήματά του και δεν μπορούμε να του αρνηθούμε καμία πληροφορία που μας ζητά. Γιατί αν ε, του αρνηθούμε ή αν ένα τμήμα του τομέα του κλάδου θεωρεί ότι πρέπει να αρνηθούμε ένα τμήμα των πληροφοριών, αν δεν παρέχουμε ένα τμήμα των πληροφοριών, αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουμε να κρύψουμε. Και να σας πω ότι εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος αν όλοι Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε στο δυνατόν περισσότερε πληροφορίε, αλλά χρειαζόμαστε και βοήθεια για να μπορέσουμε να έχουμε μία ετικέτα πολύ πιο ελεγχόμενη και μία ετικέτα που να είναι πράγματι να αποτελεί μία εγγύηση για το προϊόν που θέτουμε σε εμπορία. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζουμε το εξής. Αν αυτό είναι η Ευρώπη, αν εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι αποφάσεις ε, που θα ληφθούν να ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων του ενός και των απαιτήσεων του άλλου. Και επαιτούμε, ας απαιτήσουμε επίσης από τα προϊόντα που εισάγουμε τις ίδιες εγγύησεις όπως απαιτούμε από τα προϊόντα που εμείς αλλιεύουμε και θέτουμε σε εμπορία. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες. Ας ε, περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Στίβενσον. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις καταπληκτικές παρουσιάσεις που έκαναν. Μια πολύ σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Φερνάντες, ως προς το τελευταίο σημείο που έθιξε. Καταρχάς να του πω ότι τα αρχικά σας εισαγωγικά σχόλια για τη συμφωνία με το Μαρόκο Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι μία, από μία από τις βόρειες χώρες, αλλά ουσιαστικά υπήρχαν στην Δυτική Σαχάρα δύο σκοτσέζικα, σκοτσέζικα σκάφη. Επομένως, όταν μιλάμε για σήμανση, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κατηγορούμε τους πάντες, ορισμένοι είμαστε αθώοι. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της σήμανσης, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει ένα οικολογικό σήμα, ένα ενιαίο οικολογικό σήμα. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει κανόνες τους οποίους όλοι πρέπει να ακολουθήσουν στα πλαίσια του κλάδου της αλίας. Αν όμως θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα υψηλότερο, αν θέσει υψηλότερα τον πύχη, αν θέλετε, και θα μπορούσε ενδεχομένως ε, ένα κράτος μέλος να χρησιμοποιεί ένα οικολογικό σήμα εφόσον καταφέρει να πετύχει ένα υψηλό επίπεδο επιδόσεων, ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου, να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ευρωπαϊκό ενιαίο οικολογικό σήμα, το οποίο ενδεχομένω να μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τα πολλά διαφορετικά σήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα μπορούσε επίσης ένα τέτοιο οικολογικό σήμα να χρησιμοποιηθεί σε θελούσια βάση από αυτούς που επιθυμούν να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από εταιρείες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες και θα πρέπει να υπάγονται ακριβώς τα ίδια κριτήρια, να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με, που, με αυτές που ακαλούμεθα και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσουμε. Αν λοιπόν χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο ενιαίο σήμα, θα πρέπει οι ξένες εταιρείες να συμμορφωθούν με αυτό. Ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ κυρία so Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το πάνελ αυτό. Ήταν πολύ ενθαρρυντικά αυτά που ακούσαμε, ακούσαμε νέα στοιχεία. Θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω την κυρία Τατιάνα Γκέρλινγκ. Ε, πιστεύω ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπατε ότι το 60% των ψαριών που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγόμενα και ε, εγώ δεν ήξερα ότι τόσο μεγάλο μέρος των λευκών ψαριών ε, του Κορέγονου ε, μεταποιείται στην Κίνα. Αυτό αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία όμως όπως είπατε. Ε, την πρόκληση την δείξατε πολύ καλά στην ε, διαφάνεια σας, όπου φαίνονταν όλα τα βήματα από τα οποία περνάει ένα ψάρι όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, ότι οι διάφορες ε, αρχές πρέπει να συμπληρώσουν διάφορα έντυπα. Δεν θυμάμαι πόσα βήματα έπρεπε να περάσει το ψάρι προτού καταλήξει στο πιάτο του καταναλωτή. Εμείς είμαστε ο αδύνατος κρίκος ε, στην αλυσίδα. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βελτιώσει τα κριτήρια για ε, το πιστοποιητικό αλίας. Πόσο ε, αξιόπιστα είναι κατά τη γνώμη σας τα πιστοποιητικά Ε, Δηλαδή, έχει γίνει αλία με τρόπο βιώσιμο και νόμιμο. Ξέρω ότι υπάρχουν ιδέες όσον αφορά την ηλεκτρονική ανιχνευσιμότητα. Έχετε εξετάσει το θέμα αυτό και οι Κινέζοι παραγωγοί τι λένε. Ποιε είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτοί όταν ε, λαμβάνουν από τη Ρωσία, από την Ορβηγία όλα αυτά τα ψάρια. Οι Κινέζοι πώς ε, διασφαλίζουν ότι τα ψάρια που λαμβάνουν είναι νόμιμα. Το επόμενο βήμα είναι να τα εξάγουν σε εμά και να παρουσιάσουν και σε εμά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ομιμότητα των ψαριών. Μήπω θα μπορούσατε να, να πείτε λίγα λόγια γι' αυτό. Στον κύριο Μάρτινσον να πω ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε την ε, πρόοδο που έχει να γίνει όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα με βάση το DNA. Είμαι πεπισμένη ότι υπάρχουν πολιτικές εφαρμογές ε, για την τεχνολογία αυτή, όσον αφορά τις απάτες με αντικείμενο τα ψάρια, τα δύο είδη, τα ψάρια ιουγιού, πλά δηλαδή, ε, και ψάρια που ε, ε, αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με Ω διαφορετικά ψάρια από αυτά που είναι. Ξέρω ότι στην Ιρλανδία και στη Σκωτία έγιναν δύο διαφορετικές μελέτες όπου ψάρια που πολλούνταν ως ένα είδος ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και ε, είχαμε ε, και με άλλα ψάρια τέτοια ε, θέματα. Με την MSC όσον αφορά τον μαύρο μπακαλιάρο είχαμε επίσης ένα σκάνδαλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα, να έχουμε καλύτερη συνεργασία με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως να έχετε κι εσείς κάποιες ιδέες σχετικά με το πόσο μπορούμε να λάβουμε αυτή τη γνώση. Και στον τελευταίο μιλητή να πω ότι με εντυπωσιάζει η δουλειά σας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι μαζί θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε οι προσπάθειες σας και οι επιθυμίες ε, του καταναλωτή να συμπίπτουν τελικά. Ε, ε, ψάρια ε, ε, βιώσιμα, υγιεινά από βιώσιμη αλληλεία με τη σωστή επισήμανση. Νομίζω ότι ο καταναλωτής θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερα αν πράγματι γνωρίζει από πού προερχόνται τα ψάρια. Είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε απόλυτα και πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ακριβώς από πού προέρχονται τα ψάρια, διότι πρόκειται για άγρια ζώα. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια από τα ε, ε, αποθέματα απειλούνται και θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχονται. Κύριε Στίβενσον, ε, θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει η μεταρρύθμιση αυτή, να φροντίσουμε να υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες και πολύ καλύτερη ανιχνευσιμότητα και να έχουμε περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγα θα είμαι σύντομη, γιατί ουσιαστικά τέθηκαν ερωτήσει. Ε, θα ήθελα για να επιμείνω στο θέμα τη οικολογική ετικέτα. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, όταν ε, γνωμοδότησε για το θέμα αυτό, είπε ότι θα ήταν καλό να έχουμε μια τέτοια οικολογική ετικέτα μια τέτοια επισήμανση και συμφωνώ όμως είπατε η σύγχυση που υπάρχει τώρα στον καταναλωτή είναι μεγάλη και για το Συμβούλιο ε, επιστασίες των θαλασσών, ξέρετε, δεν δόθηκε νέο πιστοποιητικό ε, για το σολομό της Αλάσκος, γιατί ζήτησε το προϊόν αυτό να βγει από το MSC. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό το θέμα, άπαξ με μια τέτοια οικολογική επισήμανση και μετά έχουμε το πιστοποιητικό λευμάτων στον κανονισμό 1005 για την αλία πλά. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα το πιστοποιητικό, όπως είπε και η κυρία Λεβέν, έγκυται στο ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις απαιτήσει του πιστοποιητικού. Δεν ελέγχονται καθόλου τα πιστοποιητικά αυτά και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένε χώρε όπω την Παπουένα Νέα, διεξάγει έρευνα και θα ήθελα να ξέρω τι είναι, ε, ποια είναι τα αποτελέσματα γιατί ε, εγώ άκουσα ε, Παραδείγματο χάρη ε, υπαλλήλου τη Κομισιόν ε, να λένε ότι η Νέα δεν πληρεί, δεν σέβεται τις προποθέσει του πιστοποιητικού. Έτσι λοιπόν, αν τελικά δεν ελέγχονται τα θέματα αυτά, δεν σεβόμαστε τον κανονισμό 1005. Και επιμένω, ε, στον MCC τώρα πιστοποιήθηκε ο τόνος της Παππούα Νέα Γουινέα και παρόλα αυτά που λέμε άλλαξε το πιστοποιητικό για τον τόνο της Παππούα Νέας Γουινέας. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν εμπιστεύομαι καθόλου αυτές τις ιδιωτικές οντότητες. Έτσι λοιπόν, ε, κάθε φορά είμαι όλο ένα και πιο πεσμένο ότι χρειάζεται μια οικολογική ετικέτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον κάποια ελάχιστα πρότυπα για την οικολογική επισήμανση και είμαι όλο ένα και πιο πεσμένο ότι ο κανονισμός 1005 με τα πιστοποιητικά ε, για ε, τα αλλιεύματα δεν έχει καμία χρησιμότητα γιατί δεν ελέγχεται. Έτσι λοιπόν το θέμα του ελέγχου είναι δύο φορές πιο σημαντικό και Επίσης, το 45 για τις πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις επισημάνσεις σε αυτό το νέο κανονισμό φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα είναι πληροφορίε που θα μπορούν να επαληθευτούν. Γιατί τότε σε τι χρησιμεύει να έχουμε ακούσει πληροφορίε αν δεν επαληθεύονται στη συνέχεια, αν δεν ελέγχονται. Νομίζω ότι αυτέ οι ακούσει πληροφορίε που θα μπαίνουν στι ετικέτε θα πρέπει να ελέγχονται για να υπάρχει αξιοπιστία. Γιατί διαφορετικά, κοιτάξτε, κάθε φορά εγώ που βλέπω ετικέτε εξετάζομαι το μεγεθυντικό φακό και πιστεύω τα μισά. Μάλιστα να δώσω το λόγο στους ομιλητές για να απαντήσουν σημαντικά, συνοπτικά με συγχωρείτε, τόσο ακούστηκαν. Παρακαλώ. Thank you for... Σας ευχαριστώ για τις πολύ καλή ερωτήσεις που άκουσα. Θα, θα σας μιλήσω για το θέμα του πιστοποιητικού ε, ε καθώς και της Κίνας. Ε, καταρχήν όσον αφορά τα κριτήρια για την εφαρμογή του πιστοποιητικού αλίας. Ε, πράγματι είναι επαναστατικό βήμα σε όλο τον κόσμο το να εισάγουμε αυτό το σύστημα το οποίο όχι μόνο ε, είναι σημαντικό για την βιομηχανία. Χρειαζόμαστε ε, κανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες να θέσουν πρότυπα για όλο τον κόσμο και ε, αυτό θα ήθελα να αναφέρω σήμερα. Οι εμπειρίες ε, της Κίνας ε, και τα τελευταία δύο χρόνια ε, πήγα επανειλημμένα στην Κίνα και είχα συναντήσεις με τον τομέα της αλίας και των τροφίμων. Είδαμε ότι εισήχθησαν τα πιστοποιητικά αλίας, ωστόσο οι εμπειρίες τους είναι οι εξής. Δεν υπάρχει ενιαία μορφή, υπάρχουν πιστοποιητικά από διαφορετικές χώρες, έχουν διαφορετική μορφή και απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων και ποικίλουν τα πιστοποιητικά αυτά λίας. Κάποια προέρχονται από κάποιες χώρες ο, ηλεκτρονικά, άλλα, άλλα πιστοποιητικά έρχονται ε, σε χαρτί και <clears throat> θα πρέπει να θεωρηθούν και τα δύο πιστοποιητικά εξίσου έγκυρα. Αποτελεί λοιπόν ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε να θέσει ε, σαφείς κανόνες ε, που θα ε, καθορίζει πώς, ε, τι μορφή θα πρέπει να έχει το πιστοποιητικό. Και μάλιστα αυτό ξεπερνάει τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας. Η Κίνα είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα και η αρκεί να φέρει το βάρος της απόδειξης για το σύνολο της αλυσίδας της απόδειξης. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα από τη δική μας προοπτική που να προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, για να ε, διασφαλιστεί κάθε βήμα στην ε, αλυσίδα. Και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, ποιο θέει, η Κίνα φταίει. Δεν θέλω να πω ότι η Κίνα είναι τέλεια, είναι μια τεράστια αναπτυσσόμενη χώρα, χώρα έχει κάνει ε, τεράστια βήματα, είναι ανοιχτή απέναντι σε αλλαγέ, είναι ανοιχτή στο να ακούσουν τι πρέπει να αλλάξουν και γιατί. Ε, Η Κίνα εξαρτάται πάρα πολύ ε, από τις εισαγωγές και εξαγωγές ε, θαλασσινών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις όλων των αγορών με τις οποίες συνεργάζονται. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω τη τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσουν το θέμα της γιατί διότι πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή, διότι η κινέζικη βιομηχανία είναι ανοιχτή προς συζήτηση. Και επίσης μπορώ να σας πω ότι όταν πριν από δύο χρόνια συναντήθηκα για πρώτη φορά με τους μεταποιητές στην Κίνα, μου είπαν ότι η Ευρωπαϊκή ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ε, ΠΛΑ, ε, IUU δηλαδή, αποτελεί ε, εμπόδιο για το εμπόριο, ότι ο μόνος στόχος του κανονισμού αυτού ήταν να εμποδίσει την είσοδο της Κίνας στην, στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τι έκανε, βρήκε άλλους εμπορικούς εταίρους η Κίνα. Με όλα αυτά δημιουργήθηκε σύγχυση και δεν επιτεύχθη ο στόχος να γίνει πιο διαφανής η αλυσίδα προμήθειας, αλλά τα ψάρια τελικά καταλήγουν σε χώρες που δεν έχουν σύστημα ε, πιστοποιητικού ε, αλίας ε, και Γι' αυτό θα ήθελα να ενθαρρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνομιλήσει με τι ε, βασικέ ε, χώρε εξαγωγή και τι χώρε εισαγωγή, ε, την Κίνα, τη Ρωσία, τι Ηνωμένε Πολιτείε, την Ιαπωνία. Αυτέ είναι οι χώρε που καθορίζουν του κανόνε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούν λοιπόν να λυθούν τα προβλήματα αν ε, συνομιλήσουμε μαζί τους. Ε, δεν λέω ότι ε, είναι εύκολο αυτό, αλλά μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Αυτά λίγο πολύ είχα να πω όσον αφορά την παρακολούθηση, αυτά, όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Φράγα και αυτό που ανέφερε η κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ τον κύριο, στον κύριο Στίβενσον. Θα ήθελα να πω πως ε, ξέρω ότι δεν είναι ε, όλα τα ίδια και στο Νότο έχουμε κάποιες ε, εταιρείε, όπως συμβαίνει και με τον κύριο Μέιρο, ο οποίος ανέλαβε να καταψηφίσει ε, όμως ε, ξέρουμε τι κάνετε και εσείς εδώ. Αυτό είναι καλό και ενημερωνόμαστε πάντως, όπως και να έχει. Ε, νομίζω ότι και εσείς να έρθετε εκεί και να γνωρίσετε αυτή την πραγματικότητα είναι σημαντικό, γιατί αναφέρθηκε το θέμα της συμφωνίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Βασιλείου του Μαρόκου για ένα θέμα, γιατί στο Ισπανικό στόλο που δραστηριοποιείται στην επαρχία της Κάδιτ ε, έγινε λόγο για το στόλο του Κονίλ του Αλχεσίρας αλλά έχουμε και το στόλο της Ταρίφας που αλλιεύει η Λιθρίνη. Έτσι λοιπόν ε, το θέμα της Ελληνική συμφωνίας με το Μαρόκο απλώς μας δίνει μία εγγύηση ασφαλείας. Δεν ξέρω αν με κατανοείτε. Πρώτα, σας είπα πριν ότι τα στενά είναι πολύ στενά και σας είπα ότι τα ύδατα σε αυτά και, σε, και στις δύο όχθες ε, πρέπει να ψαρεύουν ε, και οι δύο στόλοι. Και εσείς ε, ξέρετε ότι... όταν δεν υπάρχει συμφωνία υπάρχει ανασφάλεια δικαίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Υπάρχει ανασφάλεια δικαίου. Και αυτό σημαίνει ότι αν δεν σκεφτείτε τη συμφωνία και ούτε η Κομισιόν ε, σκέφτεται τη συμφωνία, εγώ θα συζητούσα εξ ονόματο ε, των ελαιών των στενών του Γιβραλτάρ τουλάχιστον να σκεφτείτε μια συμφωνία γειτονία. Γιατί ε, πραγματικά υπάρχει επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, γιατί δεν θέλουμε ενισχύσει, θέλουμε μόνο να δουλέψουμε. Και αυτή η συμφωνία γειτονία θα μπορούσε να μα επιτρέψει να μπορούμε να αλλιεύουμε και στις ε, δύο πλευρές της Μεσογείου. Και αυτό που θέλω να πω σε εσά και να απαντώ και ταυτόχρονα στην κυρία Λέβεν ότι ειλικρινά εγώ πιστεύω ότι η οικολογική επισήμανση είναι κάτι θεμελιώδες. Το πρόβλημα ίσως να έγκυται στο κόστος. Κάρμεν και εσύ το ξέρεις καλά, υπάρχει πρόβλημα με όλες αυτές ε, που σου δίνουν έτσι μια ξερή ετικέτα και τελικά όλα χρήματα είναι και όλες οι συνέπειες πέφτουν πάνω στον Ελία και βρισκόμαστε τελικά στην κατάσταση να μπορούμε να υποστηρίξουμε το κόστος κανένας είδους ε, επισήμανσης. Όμως μια οικολογική ετικέτα, μια οικολογική επισήμανση θα ήταν κάτι θεμελιώδες. Εγώ τολμώ να πω και ελπίζω να μην ε, υπάρχουν αλείς που θα ε, κοιτάξουν μετά με μισό μάτι. Εγώ θα έλεγα να έχουμε υποχρεωτική τέτοια επισήμανση. Γιατί θα ήταν καλό όλοι να αλλιεύουν όπως πρέπει να αλλιεύουν με την επιλεξιμότητα, με τα επιλεκτικά εργαλεία, δηλαδή να έχουμε ένα αγκίστρι που να πιάνει τα ψάρια του μεγέθους που πρέπει ε, να αλλιεύουμε με το δίκτυ ε, που θα έχει, το οποίο το μάτι θα έχει μέγεθος ε, που θα πιάνει τα μεγάλα ψώρια. Γιατί το να διαφυλάξουμε το λευτικό πεδίο δεν είναι δεμελιώδες ε, για τους επιστήμονες, αλλά κυρίως για τους αλείς. Γιατί ένας αλλιές, ο οποίος ε, δεν είναι αυτός ο οποίος προσέχει το περιβάλλον και έχει κατά νου τη βιωσιμότητα, τελικά σκάβει το λάκκο του. ουσιαστικά καταργεί το μόνο μέσο που του επιτρέπει να φέρει ψωμί στο σπίτι του. Έτσι λοιπόν, ε, οι πρώτοι που πρέπει να το επιδιώκουν αυτό είμαστε εμείς, οι Ελλείς, κανένας άλλος. Είναι αλήθεια ότι φυσικά πρέπει να είμαστε και λογικοί και να σκεφτόμαστε ότι από την Ευρώπη και από τους οργανισμούς που δίνουν τις ενισχύσεις ε, πρέπει να δίνουν ενισχύσεις σε όποιον πρέπει, όχι σε αυτούς που μπορεί να υποσκάψουν το μέλλον. Και να μην ξεχνάμε ότι στις παράκτιες περιοχές όπου έχουμε και περισσότερη ζέστη, έχουμε ένα πρόβλημα. Η βιωσιμότητα ε, στοχεύεται μόνο προς τον ελία, αλλά όχι ε, προς την ε, αλίευση χωρίς έλεγχο. Εδώ μιλάμε πολύ συχνά για την ε, λαθρέα και άνερχη ελία, αλλά δεν αναφέρεστε στην ανεξέλεκτη αλία που γίνεται από ένα τμήμα του στόλου που δεν είναι ο στόλος ο ψυχαγωγικός, ε, ε, ούτε οι επαγγελματίες αλείς, αλλά πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που αλλιεύουν για ψυχαγωγία, αλλά με επαγγελματικά εργαλεία. Και αυτό γίνεται σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης και αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό θα συζητούσα όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα της βιωσιμότητας δεν ε, αφορά μόνο αυτούς που αλλιεύουν, αλλά και άλλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερνάντες. Μια ακόμη παρέμβαση. Yes, thank you very much for... Ο κύριος Μάρτισον, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τις προτάσεις σας. Όσον αφορά τη συνεργασία, μα προφανώς ε, θα ήθελα και εγώ να δω αν υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια συνεργασίας. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό την χρήση της γενετικής πολύ περισσότερο για στόχους ιχνηλασιμότητας. Εφόσον προκύπτει συνεχώς επίσης το ζήτημα του οικολογικού σήματος, πρέπει να σας πω ότι το Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί ένα σήμα τέτοιο για διάφορα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά. Εξετάζουν λοιπόν τα διαθέσιμα προϊόντα και για όσα προϊόντα τουλάχιστον φέρουν το δικό του σήμα, πιστοποιούν ότι προέρχονται από τις σωστές περιοχές... έχουν αλλιευθεί με τους κατάλληλους τρόπους και ούτω καθεξής Δυστυχώ όμω στι έρευνε που κάνουν δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα πορίσματα των ερευνών αυτών. Τώρα, όσον αφορά τα διάφορα συστήματα καταπολέμησης της ε, απάτησης και της ψευδούς ε, σήμανσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει ενδεχομένω να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα ζητήματα αυτά, γιατί είδαμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά, πάρα πολλοί τόνοι αλλιευμάτων που έχουν εντοπιστεί χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ε, μεθόδους αυτής. Υπήρχαν μάλιστα και διάφορες δικαστικές υποθέσεις, μερικές δικαστικές υποθέσεις εκκρεμούν ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη φυλακή ή που έχουν ε, ε, έχει χρειαστεί να καταβάλουν εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση. Πράγμα το οποίο κατατεκνεί τελικά ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, τεχνολογία DNA, τη γενετική. Να σας πω επίσης ότι στην κοινή αλληλευτική πολιτική και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 όσον αφορά την επιτήρηση. Αναφέρεται η γενετική και οι σχετικές τεχνολογίες στα ζητήματα του ελέγχου και της επιτήρησης ως προς την εφαρμογή προκύπτουν διάφορα προβλήματα και ότι ευθύνη, την ευθύνη τελικά φέρουν εν μέρη τα κράτη-μέλη και εν μέρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέγεται ότι χρειάζονται περισσότερο πιλωτικά προγράμματα. Το άρθρο αυτό είναι πολύ καλό γιατί από όσο γνωρίζω πρώτη φορά σε τόσο υψηλό νομοθετικό επίπεδο γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες αυτές στον τομέα της αλίας. Το πρόγραμμα F CP7 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από τον ε, Ευρωπαίο φορολογούμενο και πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθηθεί, να χρησιμοποιηθεί λίγο περισσότερο. Νομίζω δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν πλέον μόνο οι ερευνητέ, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε και στην πράξη. Πρόσφατα μίλησα με μέλη της ε, Ιταλικής ε, των Ιταλικών λιμενικών αρχών και είδα ότι δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να κάνουν αναλύσει, προκειμένου να ελέγξουν διάφορα προϊόντα. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα επικοινωνία και ενημέρωση και ελπίζω να καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, που ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια τη ακρόαση αν το επιθυμεί. Κύριε Ραμπού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας αφήσατε να συμμετάσχουμε. Σε σχέση με αυτά που λέγαμε όμως χθες και σε συνέχεια των όσων είπαμε χθες, νομίζω ότι ε, οι παρεμβαίνοντες ε, μας αποσαφήνισαν πάρα πολλά πράγματα. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα τώρα. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι εντελώς παράλογη για πάρα πολλούς τομείς. Νομίζω ότι σαφώς θα πρέπει να καλύψουμε ακόμα πολύ έδαφος προκειμένου να καταφέρουμε να ορίσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα, κυρίως τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών. Νομίζω όμως ότι καταφέραμε να πάρουμε συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τις προσδοκίες του κλάδου η AOP μας είπε ότι δημιουργεί μια πλατφόρμα συζητήσεων. Νομίζω ότι έχουν αποφεληθεί πολύ από αυτό. Και σαφώς υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω να πω λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Έχω καταγράψει τα όσα υπόθηκαν και κατέγραψα επίση και τι ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Στίβενσον για τα συμπεράσματα. Παρακαλώ, πολύ σύντομα, κύριε Στίβενσον. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω πάρα πολλές σημειώσεις, δέκα σελίδες σημειώσεις ε, πήρα στο λάπτοπ μου. Και αυτή είναι η πλέον πρόσφατη μια σειρά διαβουλεύσεων και που είχα με ε, πάρα πολλούς εκπροσώπους ε, στα μεγάλα έθνη που δραστηριοποιούνται στην Αλία και στις Βρυξέλλες αλλά και στα κράτη-μέλη. Αλλά χθε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση γιατί λάβαμε κάποιες νέες πληροφορίες και επίσης ε, ακούσαμε από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ε, ορισμένα από τα πιο επίμαχα σημεία που προκύπτουν με αυτή τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ, όχι μόνο για το, τα, τις και το ρόλο των ε, οργανώσεων παραγωγών, και το τι θα γίνει ε, με τους μηχανισμούς παρέμβασης ε, και για το αν ε, θα ζητήσουν να συνεχιστούν αυτοί οι μηχανισμοί παρέμβασης ή αν θα συμφωνήσουν με την προσέγγιση της Κομισιόν. Καλύτερο συντονισμός της αλίας και των εκφορτάσεων είναι κάτι που τόνισα στα έγγραφα εργασία μου και νομίζω ότι το δεύτερο τμήμα μας έδειξε και πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να βελτιώσουν όχι μόνο τον τρόπο που λειτουργούμε, αλλά και τον τρόπο που μπορούμε να διώξουμε, να ενχρώσουμε και να διώξουμε ε, όσους προσπαθούν να εξαπατήσουν το σύστημα. Η παρέμβαση περί της μοριακής τεχνολογίας ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα ε, μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που στέλνουμε και μια αντιπροσωπεία στην Κίνα για πρώτη φορά και αυτό μας ε, δίνει ε, και υλικό να συζητήσουμε με την κινέζικη κυβέρνηση να πάμε εκεί για την οικολογική επισήμανση. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα υποστήριξη για αυτά που προωθώ στο έγγραφό μου. Νομίζω ότι ήταν πολύ αξιόλογη η ακρόαση συνολικά και πάλι πρόεδρε ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που παρευρέθησαν εδώ σήμερα και μας κατέθεσαν την εμπειρία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στίβενσον. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση. Θεωρούμε ότι λίγη εδώ. Ολοκληρώθηκε και η συνεδρία της Επιτροπής Αλίας και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Θα συνεχίσει τη συνεδρία η Επιτροπή μας για να συζητήσουμε τις ελευτικές συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών. Γεια σε όλους. Καληνύχτα σας.